Uh, Καλημέρα σας. Συγγνώμη που δεν είμαστε όλοι παρόντες. Μερικοί θα έχουν κολλήσει στην κυκλοφορία, όπως και ο Επίτροπος το ίδιο έπαθε. Και έχει και πολλές δουλειές στις Βρυξέλλες βέβαια. Καλωσορίζω θερμά τον Επίτροπο Αλμούνια για την ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε. Στις 29 Νοεμβρίου ήταν η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε και θα έχουμε και άλλη μια συνάντηση στις 12 Ιουλίου. Καλωσορίζω τον Επίτροπο. Έχει πολλά να μας ανακοινώσει σήμερα. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο και μετά θα περάσουμε σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας και την Σαρμπός που με ξαναπροσκάλεσε να σας μιλήσω. Θα ασχοληθώ με θέματα σήμερα που αφορούν την ε, πολιτική ανταγωνισμό. Η εφαρμογή της κατάστασης, ε, οικονομικά συμφέροντα, αναθεώρηση των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αντιτράστ. Θα σας πω δύο λόγια για τις κρατικές ενισχύσεις για τις τράπεζες και άλλες πρωτοβουλίες μας στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα ξεκινήσουμε μια δική μας πρωτοβουλία αύριο το πρωί. Θα παρουσιάσω στους, στην Επιτροπή πρόταση για μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων και θα ξεκινήσει έτσι η πολιτική συζήτηση που μετά από μερικούς μήνες θα καταλήξει στην αναθεώρηση του πακέτου το οποίο λίγη τον Νοέμβριο. Η συνθήκη της Λισαβόνας τόνισε ιδιαίτερα τον, το, το ρόλο του τομέα των υπηρεσιών αλλά απαιτείται επίσης να διαφοροποιηθεί αυτό σε σχέση με το μοντέλο της συνθήκης και το άρθρο 6 της συνθήκης αναγνωρίζει την ανάγκη ε, καλής ποιότητας, ασφάλεια για τις ε, υπηρεσίες αυτές και ταυτόχρονα τονίζει την το ότι οι εθνικές, περιφερειακές και άλλες αρχές έχουν διακριτική ευχαίρεια στο να πώς θα οργανωθούν αυτές οι υπηρεσίες. Το άρθρο 14 ορίζει ότι η Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν αυτές οι υπηρεσίες να λειτουργούν με βάση αρχές και όρους ειδικά οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς που θα τους επιτρέπει να φέρουν σε πέρα την αποστολή τους. Και επίσης το 14 προβλέπει νέα νομική βάση για το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο και τους όρους και τις αρχές αυτές οι κρατικέ ενισχύσει δεν ισχύει για όλε τι δημόσιες υπηρεσίε. Αυτό που θα συζητήσουμε αύριο είναι μόνο για υπηρεσίε που είναι οικονομική μορφή και υπηρεσίε γενικού οικονομικού συμφέροντο. Μόνο κρατικές, κρατική χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών υπάρχει στην πολιτική ανταγωνισμού και στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Η μεταρρύθμιση που θα συζητήσουμε αύριο στην Επιτροπή στηρίζεται στις αποκλειστική αρμοδιότητα που έχει η Κομισιόν με βάση το άρθρο 106 της συνθήκης. Να ελέγξουμε τι χρήματα παίρνουν τον προπολογισμό οι υπηρεσίες αυτές. Έχουμε τη συγκυρία της κρίσης και όλο και περισσότερο στηρίζονται στις δημόσιες υπηρεσίες. Απ' την άλλη μεριά οι κυβερνήσεις χρειάζονται ρευστό. Αυτά οι δύο αντιτιθέμενες τάσεις για μεγαλύτερη ανάγκη δημοσίων υπηρεσιών και λιγότερα χρήματα στο χρηματοφυλάκιο της Ένωσης δημιουργούν μια ειδική κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει το κόστος παροχής δημόσιας υπηρεσίας είναι ένα λογικό ποσοστό κέρδους προβλέπεται, αλλά οι τρέχοντες κανόνες δεν λαμβάνουν υπόψη το πώς το κόστος αυτών των υπηρεσιών συνδυάζεται Και δεν πρέπει να πάρουμε σαν δεδομένο ότι ειδικά για τις υπηρεσίες όπου μια τέτοια εταιρεία δεν έχει επιλεγεί μέσω διαδικασίας διαγωνισμού. Είναι προς το συμφέρον της ποιότητας των υπηρεσιών και την αποδοτική χρήση των δημοσίων κονδυλίων αυτές, αυτό ειδικά για το ταχυδρομείο, για τις εταιρείες μεταφορών που έχουν μεγάλη εμπορική δραστηριότητα με κοινοτική διάσταση να ληφθεί υπόψη. Επίση, επίσης, πρέπει να διευκρινιστούν οι κανόνε έτσι ώστε οι κυβερνήσει πιο εύκολα να μπορούν να τι εφαρμόζουν και να έχουμε και νομική βεβαιότητα. Έχουμε πολλά σχόλια από όλου του ενδιαφερόμενου και από το Ευρωκοινοβούλιο έχουμε πάρει σχόλια, διότι σε μερικέ περιπτώσει παρά είναι πολύπλοκο το πακέτο αυτό. Οι νέε κατευθυντήριε γραμμέ θα λάβουν υπόψη τη μεγάλη διαφοροποίηση των υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, που έχουμε μεγάλου μεγέθου εμπορικέ επιχειρήσει μέχρι κοινωνικέ υπηρεσίε που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Παραδείγματο χάρη βοήθεια στο σπίτι για του ηλικιωμένου. Πάντω, ο έλεγχό μα θα είναι διαφοροποιημένο, πιο αναλογικό και πιο προσαρμοσμένο στη φύση των υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες για τοπικές υπηρεσίες που δέχουν μεγάλη επίπτωση στο δίκαιο του ανταγωνισμού θα απλοποιηθούν. Αύριο θα ξεκινήσει η τελική πολιτική συζήτηση. Με βάση αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε το νέο κείμενο για το νέο πακέτο το καλοκαίρι και το νέο πακέτο θα αντικαταστήσει το παλιό το Νοέμβριο. Στο μεταξύ θα σας ενημερώνω όπως έγινε μέχρι τώρα. Δεν είναι η μόνη πρόταση που έχουμε στα, στους φακέλους μας. Έχουμε ε, ειδικά πακέτα διάσωσης υπηρεσιών και αναδιάρθρωση και έχουμε επίσης και ένα πρόγραμμα για το από το 2011 και μετά για τις κρατικές ενισχύσεις για τις τράπεζες, κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις με ένα ειδικό στρατηγικό σχέδιο της Ένωσης. Αναφερούμε το καθεστώς για τα ναυπηγεία και το θαλάσσιο τομέα με την ενδιάμεση αναθεώρηση για το πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία. Όλα αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2011. Αργότερα θα ληφθούν αποφάσεις. Ξεκινάει η εσωτερική συζήτηση για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές περιφερειακών ενισχύσεων και το νέο πλαίσιο για τις επιδοτήσεις για το οπτικοκουστικά και τον κινηματογράφο επίσημη αναθεώρηση για τις κρατικές ενισχύσεις για τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες και θα ξεκινήσει και μια διαβούλευση για αυτά τον επόμενο μήνα. Μετά έχουμε την ευρύτερη μεταρρύθμιση των διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων. Οι κρατικές ενισχύσεις είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε και φέτος και του χρόνου η μεταρρύθμιση σε άλλα θέματα όπως αναθεώρηση του πακέτου των βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών αντιτράστ, ελεγκτές και οικονομικά στοιχεία που δίνει ο Chief Economist με βάση μια δημόσια διαβούλευση και εμπειρία που είχα μετά από ένα χρόνο που είμαι αρμόδιος για τα θέματα ανταγωνισμού στην Επιτροπή. Το αναθεωρημένο πακέτο θα είναι έτοιμο μετά το καλοκαίρι και έχουμε και το θέμα της συλλογικής αποζημίωσης, collective redress. Η δημόσια διαβούλευση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Απριλίου και η Κομισιόν θα εγκρίνει θέση για τις κοινέ θέσεις για συλλογική αποζημίωση επανόρθωση μέχρι το τέλος του χρόνου. Το 2012 θα προτείνω μια νομοθετική πρωτοβουλία σύμφωνα με τις αρχές αυτές. Μερικά λεπτά για το τι κάνουμε για τις χρηματοπιστωτικές εταιρείε και τις τράπεζες. Τα τελευταία χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η κρίση, χρειάστηκε να αποκατασταθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα έτσι ώστε κρίσεις σαν γι' αυτή να μην ξανασυμβούν. Ακόμα χρησιμοποιούμε το ειδικό καθεστώς για τις κρίσεις, όπως προβλέπουν οι συνθήκες. Οι συνθήκε αγορά το επιτρέπουν, γι' αυτό νέοι κανόνε διάσωση και αναδιάρθρωση των τραπεζών. Αυτό θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2012. Μου το ζητήσατε και σε μια από τις προηγούμενες συναντήσεις μας. Αναφέρθηκε μια μελέτη πώς μπορούμε να δούμε το θέμα της διάθεσης των τραπεζών. Έγινε αυτή η μελέτη και θα σας παρουσιάσω τα πορίσματα τον Ιούλιο. Όλοι ξέρετε ότι είναι μεγάλος ο λογαριασμός για το φορολογούμενο. Σας έδωσε νούμερα την προηγούμενη φορά. Δεν θα τα ξαναπώ. Το 2008 και 2009 τα κράτη-μέλη είπαν ότι χρησιμοποίησαν 2,3 δις ευρώ για τις τράπεζες. Υποστήριξη. Το 2009 1,1 δις. Για το 10 δεν έχουμε ακόμα. Θέλουμε να μείνουμε στο ελάχιστο αναγκαίο γιατί να πληρώσουν το μερίδιο τους και οι τράπεζες στη διάσωση. και να έχουν πιο υγιή και πιο βιώσιμα μοντέλα επιχειρησιακού χαρακτήρα. Επίσης, μην χρησιμοποιούνται δημόσιες ενισχύσεις για ε, να υπονομεύονται άλλοι ανταγωνιστές. Μέχρι στιγμής έχουμε 32 τέτοιες αποφάσεις διάσωσης και παρακολουθούμε από κοντά πώς οι όροι μας, αυτοί που θέσαμε, τηρούνται αν γίνεται η αναδιάρθρωση. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Έχουμε μηνύματα από την αγορά ότι μερικέ από τι επιδοτημένε τράπεζε συμπεριφέρονται επιθετικά. Όταν έχουμε απόδειξη γι' αυτό, αμέσω παρεμβαίνουμε για διόρθωση. Το κύριο πρόβλημα είναι με το που εγκρίνεται η απόφαση, δεν λύγει ο διάλογος με την Κομισιόν. Λύγει όταν είμαστε ικανοποιημένοι ότι εφαρμόστηκε η απόφαση και η τράπεζα μπορεί να στεθεί στα πόδια της χωρίς κρατική ενίσχυση και οι αποφάσεις μας να εφαρμόζονται με κάθε λεπτομέρεια. Επίσης, η αναδιάρθρωση των τραπεζών στην τράπεζα δεν έχει λήξει ακόμα. Έχουμε 24 περιπτώσεις που τρέχουν. Θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για την τελική αναδιάρθρωση τραπεζών. Και μερικές είναι δύσκολες περιπτώσεις. Είναι ο Ιρλανδέζικος τραπεζικός τομέας, όπου απαιτήθηκαν λόγω του εθνικού χρέους παρέμβαση της Ένωσης και του ΔΕΤΑΝΙΤΑΦ, τέσσερις γερμανικές περιπτώσεις του Western Bayer LD, HSH, Nordbank και Hippo Real Estate και τέλος σε μερικές περιπτώσεις στην Ελλάδα, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία. Περιμένουμε, θα περιμένουμε και κάποιες ακόμα περιπτώσεις φέτος μετά τα στρες κόπωσης. Κάθε περίπτωση αναλύεται Κάθε περίπτωση, εφαρμόζουμε όμως τις ίδιες αρχές στην αξιολόγηση. Ποιες είναι οι αρχές. Πρώτο, οι κράτες αυτές θα πρέπει να αναδιορθωθούν για να έχουν βιωσιμότητα μακρόπνοα. Πρέπει να έχουν ισχυρή κεφαλαιο, κεφαλαι, βάση κεφαλαίων, αποκατάσταση της εμπιστοσύνη τους στην αγορά, να μπορούν να δημιουργούν κέρδη για τους ε, μετόχους χωρίς να χρειάζεται να στηρίζονται σε κρατική ενίσχυση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναεστιαστούν στην κύρια δραστηριότητά του και να εγκαταλείψουν δραστηριότητα που δημιουργεί ζημιά. Δεύτερον, πρέπει να συμβάλλουν στο κόστος διάρθρωση για να μειωθεί το βάρος για το φορολογούμενο. Ο επιμερισμό του βάρους προβλέπει η, η τράπεζα να πληρώσει ένα μέρος στο κράτος για την ενίσχυα και να δίνουν μέρισμα στους ε, μετόχους μέσω κουπονιών Μόνο όταν θα υπάρχει επαρκέ κεφάλαιο στα βιβλία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τι ενισχύσει να επεκταθούν σε βάρο άλλων ανταγωνιστών που δεν έχουν πάρει ενίσχυση. Γιατί υπάρχουν πιο συνετέ τράπεζε στην Ευρώπη που δεν χρειάζεται να στραφούν στο δημόσιο πορτοφόλι υποστήριξη. Ήταν αν του επιτρέψουμε να αγοράσουν του ανταγωνιστέ με τη βοήθεια του κράτου, αυτό θα ήταν κακή πολιτική. Γι' αυτό ζητάμε οι ενισχυόμενε τράπεζε προσωρινά να μην του απαγορεύεται να αγοράσουν άλλε για να μην έχουμε στέβλωση του ανταγωνισμού, θα πρέπει οι τράπεζες να τηρούν ορισμένους κανόνες τιμολόγηση. Με δύο λόγια κάναμε και κάνουμε τη σωστή μας δουλειά ως αρχές για προστασία της δημοσιονομική σταθερότητα, των δημοσίων οικονομικών και δίκαιους και ίδιου κανόνες για όλους στην αγορά. Παράγγελα με τη δουλειά μας αυτή για την διαχείριση της κρίση ετοιμάζουμε όπως σας είπα τους μόνιμους κανόνες για την διάσωση και αναδιάρθρωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ιανουάριος 2012, αν μας το επιτρέψει η αγορά. Πάντως θα είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το νέο καθεστώς από την 1η Ιανουαρίου του 2012. Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων τώρα ως συμπλήρωμα προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη. Δύο λόγια, δύο παραδείγματα επ' αυτού. Κάρτες, πληρωμές με ίντερνετ και με κινητά. Κοιτάμε αν συνδέονται διάφορα συστήματα, αν υπάρχει προτυποποίηση, διαφάνεια. Παράλληλα με διερευνητικές πρωτοβουλίες που συζητάτε, είχαμε στιγμές προτώσεις για τη Mastercard και Visa. Οι προηγούμενες δεσμεύσεις να μειώσουν τα τέλη για διασυνοριακές πράξεις με τέτοιες κάρτες εφαρμόζονται υπό την εποπτεία ενός ε, οργάνου που έχει οριστεί. Παρόμοιες δεσμεύσεις από την Visa Europe για πιστοτικές κάρτες ε, έχουν γίνει αποδεκτές. Η έρευνά μας συνεχίζεται για τη Visa σε πιστώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα και πράξη με τις κάρτες σε νέα κράτη-μέλη. Άλλες δύο περιπτώσεις, Thomson Reuters και Standard Poor's, δείχνουν ακριβώς την προσπάθειά μας να βάλουμε σε πειθαρχία εταιρείες που είναι αναγκαίες για τον κλάδο αυτό. Με την Thomson Reuters το πρόβλημα είναι ένα κώδικα που χρησιμοποιεί για τα χρεόγραφα. Αυτοί οι κώδικες είναι αναγκαία για τους πελάτες για να μπορούν να πάρουν στοιχεία από ανταγωνιστές. Πράγμα το οποίο δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή. Αυτό θα δημιουργήσει ένα εμπόδιο που θα δημιουργήσει πρόβλημα από το να περάσει οικονομικό, από το να περάσει κάποιο από ένα πάροχο σε άλλον. Για την Standard και η περίπτωση αφορά την τιμή που χρεώνουν για, τους, ε, για τα e sings για κώδικες εντοπισμού. Έχει ένα μονοπόλιο η εταιρεία αυτή για νέα χρεόγραφα που εκδίδονται στις ΗΠΑ και εμείς θεωρούμε ότι η Standard και Poor's μπορεί να χρεώνει πολλά για την χρήση αυτών των εντοπιστών. Συγκεκριμένα, έμεση χρήστες θα πρέπει να πληρώνουν μια συνδρομή, αν και δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα για τα νούμερα αυτά. Άλλο θέμα που απαιτεί διαφάνεια και σταθερότητα για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο αναφέρεται στην λειτουργία στα credit default shops. Μέχρι στιγμής συζητάμε ποια είναι η καλύτερη λύση για μας και ελπίζω στις επόμενες εβδομάδες να μπορώ να σας αναγγείλω μερικές αποφάσεις. Άλλη εξέλιξη που πρόσφατα τράβηξε πολύ την προσοχή πολλών είναι η προτινόμενη συγχώνευση με του Euronext της Νέας Υόρκης και του Γερμανικού Χρηματιστηρίου που, αναφέρ, που αναγγέλθηκε τον προηγούμενο μήνα. Αυτή η πολύπλοκη πρόταση, deal, ε, είναι της αρμοδιότητάς μας και θα την μελετήσουμε προσεκτικά όταν θα μας το κοινοποιήσουν όλα τα στοιχεία. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και πολλά άλλα που θα μπορούσα να σας πω, αλλά χρόνο άλλο δεν έχω. Προτιμώ να σταματήσω εδώ για να περάσουμε στη συζήτηση. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ένα κατάλογο μιλητών. Θα σας το διαβάσω για να ξέρετε πότε είναι η σειρά σας. I have Jean Paul Gauzes, Andreas Schwab, Sophie Intveld, Marcus Verber, Vicky Ford, Peter Skinner. Anybody else wanting to go? Άλλος κανείς που θέλει να προσθέσουμε το όνομά του στον κατάλογο μιλητών. Όχι. Ωραία. Ο Ζαν Πολ Κοζές πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα. Πολύ πλούσια η ανακοίνωσή σας σήμερα με πολλά σχέδια θα τα ξανασυζητήσουμε, δεν σα, σας ρωτήσω για αυτά. Αλλά μια λεπτομέρεια θέλω να μου πείτε, την οποία φίξατε παρεμπιπτόντως. Είναι το θέμα των επιτροπών συναλλαγών. Θα ήθελα, μια που αναφερθήκατε στην δημοσιονομική ισορροπία των τραπεζών, να σας ρωτήσω το εξή. Οι, οι επιτροπές αυτές συναλλαγών, που καταχρηστικά μερικές φορές χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να καθορίσουν την τιμή ενός προϊόντος για πληρωμή. Ξέρετε πώς είναι οι τράπεζες, ε, πιστοτικές ή όχι, δεν θα σας τα μάθω εγώ αυτά. Αλλά τι θέτε αυτό το ζήτημα. Και θέλω να ξέρω, εσείς προβλέπετε να αλλάξετε ίσως αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί, ίσως όχι, αλλά να δείτε τι υπάρχει πίσω από αυτές τις επιτροπές ε, διασυναλλαγών και να μας πείτε αν μπορούν να καθορίσουν πραγματικά τις τιμές για τις τράπεζες. Διότι συνέπεια θα ήταν, γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει βέβαια, θα ήταν στη χειρότερη περίπτωση να κρυφτούμε πίσω από αυτές για να καθοριστούν οι τιμές έτσι ώστε το κόστος των υπηρεσιών πληρωμής να ε, αντικατοπτρίσεται σε άλλες τραπεζικές υπηρεσίες, χωρίς αυτό να γίνεται ορατό. Και βέβαια, αυτοί που δεν με πλήρωσαν βέβαια για να ρωτήσω, μου λένε ότι ίσως έτσι αυξηθεί το κόστος διαχείρισης ενός τραπεζικού λογαριασμού σε ένα μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα να το σκεφτούμε λοιπόν αυτό το ζήτημα και να δούμε αυτή η αλήθεια για τις τιμές που ψάχνετε εσείς, μήπως έχει άλλους κρυφούς στόχους και η σταθερότητα των τραπεζών πώς θα διατηρηθεί, γιατί αυτός είναι και ο στόχος. Απαντήστε ίσως χωριστά στην κάθε ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και κύριε Κοζές. Το θέμα αυτό πρέπει να το δούμε από κοντά. Από την ερώτησή σας και από αυτά που είπα εγώ, όπου αναφέρθηκα στις επιτροπές αυτές, δεν νομίζω ότι μιλάμε για ακριβώς το ίδιο θέμα. Εγώ αναφέρθηκα στις επιτροπές ε, αυτές συναλλαγών είναι το Δεμπή και Κρεντή είναι οι δύο περιπτώσεις που εξετάζουν οι επιτροπές αυτές. Υπάρχει η Mastercard που ξέρετε ότι εκεί υπήρξε μια διάκριση, χωρίστηκε και είπαμε ότι για τις debt cards θα πρέπει να είναι 0,3% ενώ για την περίπτωση των ε, άλλων να υπάρχει διάκριση. Είναι ένας υπολογισμός που κάναμε και που τον κάναμε για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάσο μερικές φορές και να μην πληρώνουμε απαραίτητα για τη συναλλαγή. Αυτό είναι κάτι που υπολογίστηκε από την Mastercard και το δέχτηκε σαν υποχρέωση και η Visa για τις κάρτες αυτές Ναι. Για τις χάρτες τις χρεωστικές είπαμε ότι κάναμε διάκριση στο ποσοστό και είπαμε ότι όλοι πρέπει να δούμε πολύ περισσότερο σε βάθος με ποιο τρόπο τελικά υπολογίζουμε το κόστος για να υπάρχει διαφάνεια. Όταν χρησιμοποιώ μια λεγόμενη χρεωστική κάρτα, debit card, για να αγοράσω κάτι, δεν ξέρω τελικά τι θα πληρώσω, τι κόστος δηλαδή θα προκαλέσω στον έμπορα που παίρνει τα χρήματά μου μέσω της πληρωμής αυτής. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Υπάρχει επίσης το κόστος για τις πληρωμές ε, το λεγόμενο direct debit, που δεν είναι και τόσο direct. Αυτό το συζητάμε και εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μέσω μιας οδηγίας που προτείνουμε εμείς. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει τέτοιο κόστος συναλλαγής. Σε πολλές χώρες υπάρχει διαφάνεια και ο χρήστης ρωτάει. Ζητάει μια υπηρεσία από την τράπεζά του και γνωρίζει το κόστος της υπηρεσίας αυτής. Και άμα δεν του κάνει, πάει σε μια άλλη τράπεζα που έχει χαμηλότερο τέτοιο κόστος. Σε ορισμένε χώρες, τις λιγότερες, δεν υπάρχει αυτή η διαφάνεια. Και δεν ξέρω τι πληρώνω σε μια τέτοια συναλλαγή όταν βάζει τέτοιο κόστος συναλλαγής μια τράπεζα, δεν με ενημερώνει. Το μαθαίνω όταν θα χρησιμοποιήσω κάποιες υπηρεσίες αυτής της συγκεκριμένης τράπεζας και όχι αν χρησιμοποιήσω κάποιες άλλες. Δεν είναι σωστό αυτό από πλευράς ανταγωνισμού, δεν είναι σωστό για το χρήστη, δεν είναι σωστό για να υπάρχει σταθερότητα. Και έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά και στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής γι' αυτό, γνωρίζοντας βέβαια ότι υπάρχει μια μειοψηφία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένε από την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Αντρέα Σφάμπ είναι ο επόμενος. Κοιτάξτε, θα βάλω το χρονόμετρο. Δεν λέω ότι πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος, αλλά όσο να είναι να ξέρει ο καθένας σας πόσο χρόνο μιλάει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε πάλι εδώ Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα της ε, ε, προστασίας της ε, ζωής σαν μια δίκαια, δίκαια μέθοδο μέτρησης. Το βρίσκω πάρα πολύ θετικό που προσπαθείτε να βρει να αξιολογήσετε τα διάφορα μοντέλα με διαφορετικό τρόπο ως υπεύθυνος για τον αγωνισμό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θέλουμε να έχουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά και δεν επιτρέπεται να ε, οπισθοχωρήσουν ορισμένες χώρες ε, όσον αφορά τον ελεύθερο ανταγωνισμό επειδή υπάρχει ιδιαίτερη υποστήριξη από το εκάστο κράτος. Κατά δεύτερον, όσον αφορά το θέμα του ανταγωνισμού. Είδατε ότι η Επιτροπή μας ε, εγκαθίδρυσε μία task force για την πολιτική ανταγωνισμού. Θα ήταν καλό να έχουμε συνεννόηση μεταξύ μας, Ιδίω γιατί όσον αφορά την ενίσχυση έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού που θα υποβάλλεται προσεχώ, θα μπορούσαν ίσως ορισμένα θέματα να αντιμετωπιστούν πιο δομημένα από ό,τι στο παρελθόν. Το πιο σημαντικό θέμα που στο πέρα αναφέρθηκε είναι το λεγόμενο collective redress. Ε, είναι σημαντικό να μπορούν ε, η Κομισιόν να αποζημιώσει τους ε, καταναλωτές που έχουν χάσει από την συμπεριφορά κάποιων επενδυτικών εταιριών και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε υπάρχει από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Δικαιοσύνης η Κομισιόν ε, να προβλέψει, να δώσει στα θύματα αυτά ένα, ένα, μια αποζημίωση κατόπιν όμως που θα έχει πρώτα κάνει μια έρευνα για να δει ε, τι γίνεται ε, σχετικά πόσο ήταν δηλαδή, πόσο έχουν ζημιωθεί κατά μέσο όρο. Θα ήταν καλό να μας απαντήσετε και στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Εννοείται ότι η πρόθεσή μας είναι κάθε είδους τρέβλωση να την καταργήσουμε. Και είμαι βέβαιος ότι με τις προτάσεις, με τις ιδέες με τις οποίες θα έρθει το Σώμα των Επιτρόπων μέσα στους επόμενους μήνες, θα έχουμε μια ακόμα πολιτική συζήτηση πριν συντάξουμε τις τελικές προτάσεις προς απόφαση και το τελικό πλαίσιο που θα αντικαταστήσει το πακέτο του 2005. Ε, λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει καμία στρέβλωση στις αγορές, κάθε άλλο η απόφασή μας, το πακέτο για τις κρατικές ενισχύσεις προς τις κοινοφελείς, ε, προς τις κοινοφελείς υπηρεσίες οικονομικού χαρακτήρα είναι κάτι που θα βοηθήσει να μην υπάρχουν τέτοιες τρευλώσεις. Και αυτό θα γίνει μέσα από διάφορες πτυχές. Έχω επιμείνει και θα το ξαναπώ σε δύο πράγματα, τα οποία εξάλλου στήριξαν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στις διαβουλεύσεις και στις συζητήσεις που είχαμε μέχρι τώρα. Πρώτον, απλοποίηση, απλούστευση του συστήματος για όλες τις υπηρεσίες τοπικού χαρακτήρα. Υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα συνήθως, που δεν υπάρχει λόγος να έχουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να είναι περίπλοκο. Πρώτα απ' όλα γιατί πρόκειται για υπηρεσίες ε, χαμηλής κλίμακας που δεν θα επηρεάσουν τόσο πολύ σημαντικά στις περισσότερες περιπτώσεις τις συναλλαγές που γίνονται στην εσωτερική αγορά, το κοινοτικό εμπόριο. Και από την άλλη μεριά δεν είναι και σε θέση να έχουν ε, χωριστά μια λογιστική απόδοση. Οπότε πρέπει να ξέρετε ότι είχαμε πάρα πολλά σχόλια προς αυτή την κατεύθυνση και έχω την εντύπωση ότι ακριβώ επειδή είναι περίπλοκο το τρέχον πλαίσιο και δεν λαμβάνει υπόψη το πόσο διαφορετικές είναι οι υπηρεσίες αυτές ολόκληρη την Ευρώπη, τελικά υπάρχει ένα τμήμα των υπηρεσιών αυτών που αγνοούμε πλήρως, που δεν τις λαμβάνουμε υπόψη στο τρέχον πλαίσιο. Γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε ένα πλαίσιο με απλοποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία που έχουν οι κοινοφελείς υπηρεσίες και να πετύχουμε αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει και που είναι οι υπηρεσίες οι οποίες παίρνουν κρατικές ενισχύσεις και που έχουν όμως τέτοια διάσταση που μπορεί να δημιουργήσει στρεβλώσει στην εσωτερική αγορά εξαιτία ακριβώ τη κρατική ενίσχυση. Προσπαθούμε να δούμε λοιπόν πώ θα βελτιώσουμε την ε, ανάλυση μα για να δούμε η αντιστάθμιση πρέπει να υπάρχει για τις υπηρεσίες εκείνες που περιλαμβάνονται στο πακέτο του 2005. Συγχρόνως, όμως, για να κάνουμε την ανάλυση αυτή, είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο για μας που είμαστε υπεύθυνοι να ελέγχουμε τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά είναι σημαντικό και για τους πολίτες. Αν ένα συγκεκριμένος ε, διαχειριστής κοινοφιλούς υπηρεσίας παίρνει ε, κρατική ενίσχυση, εννοείται ότι και πρέπει να μας δώσει το λογαριασμό, αλλά και πρέπει να διασφαλίσει ότι θα είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό στη δουλειά του. Δηλαδή, το δημόσιο χρήμα πρέπει να συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Και αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως βέβαια για τους πιο μεγάλους παροχής ε, κοινοφελών υπηρεσιών, για να μην υπάρχει ακριβώς τρέβλωση στην αγορά. Οπότε, από αυτού συμφωνούμε. Δεύτερον, έμαθα ότι δημιουργήθηκε αυτή η task force ε, για τον ανταγωνισμό. Εντάξει, πολύ χαίρομαι. Βεβαίως και να συναντηθώ ε, μαζί τους για να συζητήσουμε, να δούμε και πώς θα συνεργαστούμε. Και αυτό όχι μόνο εν ώψη της επόμενης έκθεσης για τον ανταγωνισμό, αλλά και επειδή υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες. Σε ορισμένες αναφέρθηκα, αλλά δεν τις ανέφερα όλες. Πρωτοβουλίες λοιπόν οι οποίες σιγά σιγά αναπτύσσονται. Ανεξάρτητα πάντως με το ποιος θα πάρει την απόφαση και τις περισσότερες φορές υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ξέρετε ότι θέλω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στον προβληματισμό μας και στις συζητήσεις μας για να ετοιμάσουμε καλά όλο αυτό το σύνολο πρωτοβουλειών. Και όσον αφορά τις συλλογικέ προσφυγές πρέπει να ξέρετε ότι αυτή την εποχή ε, συζητάμε τους οριζόντιους μηχανισμούς ή μάλλον πιο σωστά αρχές, τις οριζόντιες αρχές για θέματα προστασίας του καταναλωτή, περιβάλλον κλπ. κλπ. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σας, είμαστε τρεις, η Ρέντινγκ, ο Ντάβιτ και εγώ, που ε, ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα στην Κομισιόν. Στα τέλη της χρονιάς, αφού έχουμε αναλύσει τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, θα καταλήξουμε σε απόφαση. Και βάσει της απόφασης αυτής θα συζητήσουμε και θα συζητήσω Ευχαριστώ μαζί σας τις αρχές πάνω στις οποίες θα βασιστεί η νέα νομοθετική μας πρωτοβουλία για την ιδιωτική πρωτοβουλία και τι αρχές θα περιλαμβάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τη σοφή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Και θα μπορέσω να συμφωνήσω με όλα αυτά που ελέγχθησαν από τον συνάδελφο Σβάπ, αλλά θα ήθελα κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν, όταν απαντήσατε στην ερώτηση του κυρίου Γκοζέτ για το τέλος συναλλαγής, δεν ξέρω, εγώ υπέβαλα μια κοινοβουλευτική επερώτηση όσον αφορά αυτό το θέμα της ε, κακής χρήσης των καρτών και απαντήσατε ότι δεν είσαστε επεπισμένος ότι οι εξελίξεις στον τομέα δεν προχωράνε αρκετά γλίγορα ούτως ώστε να υπάρξει μια πραγματική αγορά. Δίνετε την εντύπωση ότι σκεφτόσασταν να υιοθετήσετε ε, κάποια νομοθετικά μέτρα σχετικά. Εξακολουθεί να ισχύει ή τώρα σε την εξελίσσει είναι αρκετά γρήγορε. Δεύτερον, όσον αφορά την αναθεώρηση του, της δέσμης μόρτικρους. Δεν ξέρω κατά πόσον ε, θέλουμε να υποβάλουμε εμείς προτάσεις που θα οδηγούσουν σε στρέβλες στον νομισμό, προφανώς όχι. Αλλά η πίεση η χρονική είναι πάρα πολύ μεγάλη και όταν εκφράστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2005 πάνω στη θέσμη αυτή, ζητήσαμε ευρία αξιολόγηση μετά από κάποια χρόνια. Δεν θυμάμαι να ήταν μια τέτοια αξιολόγηση. Μήπως όμως αυτό δεν θα πρέπει να ήταν η βάση για νέες προτάσεις και όχι η πολιτική συζήτηση. Πρώτα δηλαδή να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις της σημερινής δέσμης προτού υποβληθούν νέες προτάσεις. Και πάνω σε αυτό θεωρώ ότι ε, στην, στο ψήφισμα αναφέρονται ιδιαίτερα οι κοινοφελείς υπηρεσίες και δεν μου φαίνεται είναι σωστό ότι δεν είχε εμπλεκεί η δική μας Επιτροπή περισσότερο. Και τέλος, όσον αφορά την Task Force ε, για τον ανταγωνισμό που αναφέρθηκε ήδη και την πρόθεσή σας να συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε αυτά. Χαίρομαι που το άκουσα και είμαι πεπισμένη ότι η δημιουργία αυτής της Task Force θα βελτιώσει τη συνεργασία μας γιατί τα πρόσφατα χρόνια κάθε χρόνο υιοθετούμε ένα ψήφισμα με συστάσει, με σχόλια, με απαιτήσει. Έχουμε μια απάντηση από την Κομισιόν, αλλά δεν δίνει τη συνέχεια. Και ελπίζω, αν μπορούσαμε να συνεργαστούμε με στα πλαίσια αυτής της Task Force, θα πάνε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ιντφέλτ. Καταρχήν, όσον αφορά το θέμα αυτό τον γλωστικών και πιστοτικών κρατών. Κατά βάση υπάρχει ένα δύο πόλιο ε, κάτω από πολλές πτυχές. Όχι παντού, αλλά have cross uh, conversations. I uh, am following. Αλλά κοιτάξτε, παρακολουθώ νέε πρωτοβουλίε για νέε εισόδου σε την αγορά. Ε, δεν μπορώ να είμαι πολύ σίγουρος γιατί εξαρτάται από τη δυνατότητα νέας εισόδου στην αγορά. Εάν βλέπω να υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο, θα αντιδράσω αμέσω από σκοπιά ανταγωνισμού βέβαια. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, δεν μπορώ να εισαγάγω εγώ οτιδήποτε σε αυτό το τομέα. αν βλέπω κάπου που προσπαθούν να μπουν στην αγορά, θα είμαι πολύ ευτυχή να πετύχουν. Ωραία. Διακανονισμό για τα μυφ και άλλα τέλη συναλλαγή. Μίλησα με τον κύριο Κοζές όσον αφορά την άμεση πίστοση. Υπάρχει διακανονισμός εκεί. Όσον αφορά τώρα τις πιστοτικές χρεωστικές κάρτες, δεν υπάρχει διακανονισμός μέχρι στιγμής. Στη ΣΥΠΑ, ναι. Έχουν εισαγάγει κάποια διατάξεις τα τελευταία χρόνια νέους κανονισμούς για τα μυφ των καρτών. Διάβαζα ένα άρθρο στον τύπο, στον Αμερικανικό τύπο πρόσφατα, πολύ κριτικό όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτών των διακανονισμών. Που έχουν επιπτώσεις όσον αφορά τους χρήστες. Εγώ έχω πάντα αυτό το ερωτηματικό στη δική μου ανάλυση. Εγώ χρησιμοποιώ τα μέσα που έχω στα χέρια μου, αντιτράστ, ε, ανταγωνισμός, αλλά έχω, έχω ένα ερωτηματικό κατά νου. Τι θα γίνει εάν τελικά καταλήξουμε σε διακανονισμό των πιστοτικών και χρεωστικών κρατών. Δεν μπορώ να σας δώσω μια τελική απάντηση σε αυτά. Αλλά είναι ένα θέμα που το έχω πάντα κατά νου. Εστιάζει. Τώρα βέβαια προετοιμάσαμε μία έκθεση ε, αξιολόγησης που θα την οθετήσει αύριο η Κομισιόν. Το ξέχασα να σας το πω εισαγωγικά. Κάναμε όμως ε, μία αξιολόγηση με τις απόψεις των ε, κρατών μελών, των ενδιαφερομένων, τις δικές μας εμπειρίες από το 2005 και προετοιμάσαμε μία έκθεση αξιολόγησης που θα συνοδεύσει την ε, ανακοίνωση που θα αύριο. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να μπορέσω να συνεργαστώ στενά με αυτή την task force που δημιουργήσετε και αν και η Επιτροπή Απασχόληση θέλει να συμμετάσχει σε συζητήσει αυτές, θα είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής να συζητάω τα θέματα μαζί σα. Χρειάζεται νομίζω και μ' αρέσει κιόλα. Λοιπόν, εάν θεωρήσετε ό,τι θέλετε να συζητήσετε με μένα άμεσα ή με τις υπηρεσίες μου άλλα θέματα, να μου το πείτε. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχεί κάθε φορά που μπορούμε να έχουμε το διάλογο αυτό μαζί σα. Αλλά όμως υπάρχει ένα αλλά. Διάλογος, ανταλλαγή απόψεων, συζητήσεων δεν σημαίνει ότι ε, τα θέματα αυτά για τα οποία είσαστε εσεί πλήρως υπεύθυνοι θα προσπαθήσω να επιβάλλω δική μου άποψη. Και από την άλλη μεριά βέβαια διάλογο πάλι δεν σημαίνει ότι για το θέμα για το οποίο εγώ η Κομισιόν είναι πλήρη υπεύθυνη θα επιβάλλετε τη δική σα άποψη. Θα ακούσουμε προσεκτικά, θα συζητήσουμε τα επιχειρήματα, θα ανταλλάξουμε απόψει και μετά στι 90% των περιπτώσεων θα συμφωνήσουμε, είμαι σίγουρο. Αλλά τι θα γίνει με το άλλο 10% πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Πρόεδρος, θα προσπαθήσουμε, αλλιώς δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε, λέει πρόεδρος. Πίτερ Σκίνερ είναι στην Task Force και μετά θα επανέλθω στον Μάρκος και τη Βίκη. Θα σύντομο. Μία υπόδειξη. Καταρχήν συγχαρητήρια γιατί για τότε ασχοληθήκατε με τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην Task Force. Μία υπόδειξη. Το δεν υπάρχει διαφάνεια δεν το θεωρείτε σημαντικό για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Αναφερθήκατε στα διαδικασία των στρες κόπωσης, το, συγγνώμη, των τεστ κόπωσης. Καλό θα είναι να φροντίσουμε από κοινού να γίνουν σωστά. Επίσης, δεν θα μπορούσατε να κοιτάξετε και άλλες δομές στην τράπεζα, παραδείγματος χάρη για τα ταμιευτήρια στην, τράπεζα, στην Ευρώπη, που είχαν ε, ωφέλη κακώς Βέβαια δεν έχουν σχέση με την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά έχουν κάποια σχέση. Αναφερθήκατε στο γερμανικό χρηματιστήριο και τις χρηματιστήριες της Νέας Υόρκης. Πρέπει να το δείτε το θέμα αυτό, όπως επίσης και την νομοθεσία τη σχετική που συζητάμε εδώ. Πρέπει χάρη για, για τα παράγωγα. Έχουν σχέση όλα αυτά μεταξύ τους, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Σκίνερ. Συμφωνώ ότι χρειάζεται διαφάνεια. η διαφάνεια είναι πάντα καλή. Ιδιαίτερα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εμείς ως νομοθέτης έχουμε πολλή δουλειά. Βέβαια, εσείς και το Συμβούλιο τελικά θα επιβάλλετε το πώς και πόση διαφάνεια θα μας βοηθήσει να έχουμε πιο υγιή και φερέγγια ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να προστατεύονται και οι πελάτες τους. Γιατί η έλλειψη διαφάνειας είναι και κίνδυνος όσον αφορά τον ανταγωνισμό αλλά και μεγάλος κίνδυνος για την σταθερότητα όπως διδαχτήκαμε από την κρίση. Ελπίζω τα τεστ κόμπωσης που θα γίνουν σύντομα θα είναι επιτυχή. Δεν συμφωνώ ότι ότι έχουν πλεονεκτήματα τα, τα Γενικά. Αυτό αξίζει να συζητηθεί αν έχουν κάποιο ειδικό πλεονέκτημα ή όχι. Έχουμε διαφορετικά νομικά αρχιτεκτονήματα για τα χρηματοπιστωτικά εδρήματα. Πρέπει όμως να επιπτεύω, εποπτεύονται να διέπονται από τον ίδιο κανονισμό όσον αφορά την συνετή διαχείριση, τη σταθερότητα του συστήματος κλπ. Μία περίπτωση που την ξέρω καλά, τις, ε, τα ισπανικά τα ταμιευτήρια, αυτό συμβαίνει. Μερικές τέτοιες ε, τράπεζες τέτοιου είδους καταθέσεων, τα προβλήματά τους δεν έχουν σχέση με κακή εποπτεία. Έχουν σχέση με την στεγαστική φούσκα. Αυτή οδήγησε στο να μην υπάρχει εποπτεία μακρο ε, χρόνιου χαρακτήρα και δημιουργήθηκε ένας συστημικός κίνδυνος. Δεν υπήρχε τέτοιου, τέτοιου είδους ε, μακρόπνοη ε, εποπτεία. Και αυτό ήταν ένα από τα κύρια κενά όσον αφορά την υποδομή, την εποπτική υποδομή. Συμφωνώ με το τρίτο σχόλιο σας συγχώνευση γερμανικού και αμερικάνικου της Νέας Υόρκης χρηματιστηρίου επιθυμίου που θα μας κοινοποιήσουν τον deal. Μέχρι στιγμής είχαμε μερικές πρώτες επαφές, ακόμα επίσημα δεν μας κοινοποίησαν τίποτα. Θα αναλύσουμε αυτή τη συγχώνευση αλλά πρέπει να συντονιστούμε με σας και στο Συμβούλιο που συζητάτε νομοθεσία για τα παράγωγα και την πρωτοβουλία του ΕΜΗ. Γιατί το, το Γερμανικό Χρηματιστήριο και το New York Euronext με τα παράγωγα στηρίζονται πάρα πολύ στενά. Άρα θα το συζητήσουμε με εσάς. Πρόεδρος, Συνεχίζουμε με τον Μάρκο Φέρμπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δίνετε το λόγο στους συναδέλφους χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια. Γιατί εντάξει, εσείς αποφασίσετε σε μια ποια θα μιλήσουμε, αλλά δεν μου άρεσε πάρα πολύ Μου με πήρατε προς τα πίσω. Κύριε Επιτροπή, αναφερθήκατε στην αξιολόγηση των ε, κρατικών ενισχύσεων για τις τράπεζες. Εσείς αναφερθήκατε γενικά στις Ιρλανδικές τράπεζες και τις τέσσερις τράπεζες στην ε, Γερμανία, εκ των οποίων οι τέσσερις ε, ανήκουν σε ομοσπονδιακά κρατήδια. Δεν ξέρω κατά πόσον η Κομισιόν, όπως είπατε εσείς, πραγματικά χρησιμοποιεί τα ίδια μέτρα και τα σταθμά, γιατί μια χώρα όπως η Ιρλανδία που δεν ήθελε, αρνήθηκε στην αρχή να κάνει μια αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των τραπεζών και οδηγήθηκε στο χείλος του γκρεμού και θα πληρώσουν τώρα οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πρέπει να αξιολογηθεί διαφορετικά από μια τράπεζα η οποία πάντα είχε διαφορετική δομή και χρηματοδοτεί το πάντα από το κράτος. Δηλαδή οι, οι τράπεζες που ανήκουν στα ομοσπονδιακά κρατήδια. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα λειτουργούν τραπεζικό σύστημα σε ορισμένα κράτη-μέλη που να λαμβάνει υπόψη όλες τις διαφορετικές πτυχές στη λειτουργία τους και είναι πραγματικά ε, ακατανόητο γιατί μια χώρα όπου ε, για μια χώρα πρέπει όπως η Ιρλανδία να ε, συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες ως φορολογούμενοι γιατί το κράτος έδωσε μια χωρίς όρια εγγύηση για τις τράπεζες αυτές, ενώ από την άλλη μεριά κατά βάση υγιείς τράπεζες ε, όπως τη Γερμανία δεν μετρώνται σωστά, δεν λαμβάνονται σωστά υπόψη, μετρώνται με τα ίδια σταθμά και οδηγούν στο χείλο του κρεμού και αυτές. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω καταλάβει καλά αυτό που λέτε. Θα προσπαθήσω όμως να σας απαντήσω αν κατάλαβα καλά τελικά. Αρχικά μίλησα για τις αρχές πάνω στις οποίες προσπαθούμε να προχωρήσουμε στον ε, έλεγχο των ε, ενωτήτων αυτών μετά την κρίση. Και έχουμε ένα τεράστιο κατάλογο τραπεζών. Είπα στην αρχή ότι έχουν ήδη ληφθεί πολλές ε, αποφάσεις και άλλες ξεκινάνε τώρα και τις παρακολουθούμε. Αποφάσεις που έχουν να κάνουν, δεν θα τις πω βέβαια, που έχουν να κάνουν με μεγάλες βρετανικές τράπεζες οι οποίες χρειάστηκε να δώσουν σχέδια αναδιάρθρωσης ήδη από το 2009 και υποτίθενται σε εφαρμογή με επενδύσεις, με ισολογισμούς, με αλλαγές ε, μεγαλύτερες ή μικρότερες όσον αφορά την λειτουργία τους και έχουν να κάνουν και με την συμμετοχή του κράτους με χρήματα δηλαδή που έδωσε η Μεγάλη Βρετανία. ελήφθησαν αποφάσεις και εδώ στο Βέλγιο για τις τρεις μεγάλες τράπεζες, τις Βέλγικες και στην Ολλανδία, για πολλές από τις μεγάλες Ολλανδικές τράπεζες, με δικιά μας παρέμβαση και στη Γερμανία, κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πολύ μεγάλο όπως είναι η Commerzbank ή όπως είναι η Landesbank, όπου υπάρχουν και εκεί και έχουν ξεκινήσει σχέδια αναδιάρθρωσης. Το δρόμος, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, νομίζω ότι είναι 8, όπου τελικά πτώχευσαν. Η Σάξεν έλβε και μπήκαν σε άλλη τράπεζα. Το ενεργητικό τους. Και σε άλλες περιπτώσεις είχαμε πτώχευση και στην Ισπανία δύο ε, αποταμίευσεις, τη Σουρ και της Δελαμάντσα όπου το ενεργητικό τους πέρασε σε άλλες αποταμιευτικές ε, τράπεζες. Η δουλειά λοιπόν έχει γίνει. Έχουν ληφθεί αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες έπρεπε να λάβουν υπόψη το μοντέλο λειτουργίας έτσι ώστε να ξέρουμε ότι η αναδιάρθρωση θα οδηγήσει σε έναν βιώσιμο φορέα. Μείωση όσο γίνεται περισσότερο της τρέβλωσης επειδή δόθηκαν χρήματα από το κράτος και το bank sharing ανάμεσα στους μετόχους τις διάφορες πλευρές ε, του χρηματοπιστωτικού αυτού ιδρύματος με το κράτος που έδωσε τα χρήματα. Αυτή λοιπόν ε, η διαδικασία βάσει των ίδιων αρχών που έχουν γραφτεί σε τέσσερα συγκεκριμένα κείμενα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το φθινόπωρο του 2008 μέχρι τα μέσα του 2009, αυτές οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται τώρα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκεί όπου δεν καταφέραμε ακόμα να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, όπου δεν ελήφθη τέτοια απόφαση. Πρόκειται για την περίπτωση της Ιρλανδίας, δεν είναι βέβαια όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ίδια κατάσταση. Βρίσκονται υπό πτώχευση πάντως δύο. Η Ιρλανδική τράπεζα περνάει από αναδιάρθρωση και στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και άλλες τράπεζες, τέσσερις στη Γερμανία μεταξύ άλλων. Συζητάμε λοιπόν με όλους αυτούς και ξεκινάμε από τις δικές τους ιδιαιτερότητες, γιατί το κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Και συγχρόνως δικιά μας ευθύνη είναι να θέσουμε σε εφαρμογή τις ίδιες αρχές και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξουν στρεβλώσεις ή τέλος πάντων οι στρεβλώσεις αυτές να είναι οι ελάχιστες δυνατό. Συμφωνώ με την ανάλυση πάντως που κάνετε όπου συγκρίνετε την κατάσταση των γερμανικών με τις Ιρλανδικές τράπεζες. Έχετε δίκιο για πολλού λόγου. μάλλον αν θέλετε σε κάποια άλλη συνάντηση να μπω σε λεπτομέρειες αλλά και κλεισμένο το θυρών. Πάντως δεν συμφωνώ με την ανάλυση εκείνη που λέει ότι πληρώνουμε την Ιρλανδία και γιατί να κάνουμε παραπάνω προσπάθειες από αυτές που χρειάζονται για τη Γερμανία, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή μια τέτοια ανάλυση. Η δίκη. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αλλά έχω πολλές ερωτήσεις. Θα μπορούσατε πιο συγκεκριμένα να μας μιλήσατε για τον Deutsche για την κατάσταση εκεί. Για το χρονοδιάγραμμα. Ξέρω ότι περιμένετε, αλλά ένα, ένα μήνα τώρα ανακοινώθηκε η συναλλαγή και ο χρόνος περνάει. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε περισσότερα πού βρισκόμαστε, σε ποια διαδικασία βρίσκεστε και πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Για τις Ιλλανδικές τράπεζες τώρα θέλω να ρωτήσω κι εγώ. Ακούω φωνές που λένε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δίνουμε περισσότερα χρήματα στην AB, για παράδειγμα στην BI, και θέλουμε να δούμε και οι ε, πιστωτές να αναλαμβάνουν κάποιο βάρος. Αλλά από την άλλη μεριά οι επιπτώσεις μπορεί να είναι μεγάλες σε άλλες χώρες μέλη. Μπορείτε να σχολιάσετε σε αυτά. Και τελικά για τον έλεγχο κυρίως θέλω να σας ρωτήσω. Έχουμε ελέγχους που επικεντρώνονται σε διάφορες ε, τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εμείς θέλουμε περισσότερο ανταγωνισμό όπως ξέρετε και περιμένουμε και την ανακοίνωσή σας για τον έλεγχο. Ορισμένοι λένε ότι για να ενθαρρύνουμε τον ανταγωνισμό θα πρέπει να υπάρχει εκ περιτροπής υποχρεωτικά αλλαγή στον έλεγχο. Σε χώρες μέλη όμως που αυτό συμβαίνει, οι επιχειρήσεις δεν θέλουν να περάσουν σε ένα μικρότερο έλεγχο λέτε να γίνεται εκ Αν γίνει εκ κάποια στιγμή θα υπάρχει Λιγότερο έλεγχο, περισσότερο έλεγχο Λοιπόν, δεν κινδυνεύει να χειροτερέψει η κατάσταση αντί να βελτιωθεί με ένα τέτοιο τρόπο, εκ αλλαγή στον έλεγχο. Αλμούνια, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να προκαταλάβω και να σας πω πότε δύο ιδιωτικές ε, επιχειρήσεις θα αποφασίσουν να κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συγχωνεύονται. Δικό του θέμα είναι αυτό. Δεν μπορώ εγώ να το προκαταλάβω. Όταν το αποφασίσουν εκείνοι, εκείνοι θα το έχουν αποφασίσει, δεν το έχω αποφασίσει εγώ. Όπως ε, σας ε, έχω ξαναπεί, έχω πάρει πληροφορίες και από τις δύο πλευρές για την πρόθεσή τους. Είναι μια γενική πληροφορία που έχω, όπως διαβάζουμε στα μέσα ενημέρωσης. Συναντήθηκα και με τις δύο πλευρές μου ζήτησαν να βρεθούμε προκαταρτικά, ώστε προφορικά να με ενημερώσουν και οι δύο πλευρές, οι εκπρόσωποι δηλαδή και της Euronext και της German Bolsa μου είπαν ότι εν ευθέτω χρόνο θα έρθουμε να σας δούμε, τέλος πάντων θα έρθουμε στην γενική σας διεύθυνση με την επίσημη κοινοποίηση. Αλλά πότε ακριβώς θα το κάνουν αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω, γιατί δεν είναι δικιά μου προσωπική γνώμη, είναι δικιά τους, ότι όταν γίνει η κοινοποίηση, όταν γίνει η ανάλυση, δεν θα είναι απλή μετά. Δεν θα είναι απλό να αναλύσουμε δηλαδή την κοινοποίηση για συγχώνευση. Υπάρχουν προθεσμίες και πρέπει να δούμε πώς θα τηρηθούν. Δεν θα με εκπλήξει αν η συγχώνευση αυτή άπαξ και κοινοποιηθεί δεν θα με εκπλήξει λοιπόν αν αποτελέσει μια περίπτωση η οποία θα μας αναγκάσει να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο. Αλλά όλα αυτά δεν μπορώ να σας τα πω με σιγουριά, αν δεν πάρω την κοινοποίηση δεν μπορώ να σας πω τίποτα ουσιαστικά. Τώρα για την ερώτηση που κάνατε όσον αφορά τις Ιρλανδικές τράπεζες. Αναλύουμε την κατάσταση σε αυτές. Αλλά δουλεύουμε και μέσα στην Τρόικα και είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τις Ιρλανδικές Αρχές για την εφαρμογή του προγράμματος του που αποφάσισαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνέ Μασματικό Ταμείο. Να δούμε κατά πόσο οι προποθέσει αυτές προχωράνε. Τώρα συζητιούνται με την νέα Ιρλανδική κυβέρνηση. Δεν ξέρω την Παρασκευή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τι θα πει γι' αυτά. Παρακολουθούμε πάντως στενά τις συζητήσεις. Γιατί μέρο των συζητήσεων αυτών θα έχουν συνέπειες και στα προγράμματα αναδιάρθρωσης που εμείς ε, συζητάμε. Έχουμε πρώτε επαφέ με τον κύριο Νούναν, που είναι ο νέο Υπουργό Οικονομικών τη Ιρλανδία, και του λέμε: Εσεί θα μα πείτε πότε θα είσαστε έτοιμοι να έρθετε και να μα δείτε με νέα στοιχεία. Αλλά φαντάζομαι ότι πριν από αυτό δεν μπορείς να ασχοληθείς με συγκεκριμένες περιπτώσεις, με συγκεκριμένες ε, προτάσεις. Πρώτα πρέπει να δεις το γενικό πρόγραμμα που θα έχει συμφωνηθεί ε, με την Τρόικα. Το τρίτο τώρα που με ρωτήσατε για τους ελέγχους. Είναι ένα θέμα ρύθμισης. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μπαρνιέ, ανακοίνωσε ήδη κάποιες ε, ρυθμιστικές πρωτοβουλίες για ελεγκτικές εταιρείε. Είναι νομίζω διαβούλευση. Ξεκίνησε πριν από μήνες τέλο πάντων και εμείς συμφωνούμε βεβαίως μαζί του και εγώ συμφωνώ μαζί του για το ότι όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μεγάλων παικτών Ακολουθώντας την ρυθμιστική πτυχή του ζητήματος αυτού, η εκπεριτροπής έλεγχος που λέτε είναι θέμα ρύθμισης, δεν είναι θέμα που αποφασίζουν οι αρχές επί του ανταγωνισμού. Αν πάντως κάποια στιγμή διαπιστώσω ότι υπάρχουν επιτυχίες οι οποίες απαιτούν παρέμβαση από τη δικιά μας την οπτική γωνία, από τη δικιά μας την πλευρά του ανταγωνισμού, τότε θα παρέμβω. Προς το παρόν πάντως δεν είναι θέμα φραγμών στην είσοδο. Είναι θέμα ρύθμισης που μπορεί να βελτιωθεί και πρέπει να βελτιωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω τον εαυτό μου και έχουμε 34. Νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να κάνω επίσης κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να επανέλθουμε στο θέμα της ένωσης της με την Deutsche Boss. Δηλαδή όσον αφορά το θέμα του συσχετισμού μεταξύ των καθαρίσεων και των ε, ε χρηματιστηρίων ε, ιστορικά από όσο ξέρω τα, κρατη, τα ταμεία των κρατών έχουν απαγορεύσει κάποιες κινήσεις ε, σαν αυτές που προτείνονται τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό σχετίζεται και με το διεθνές περιβάλλον και το θέμα του αναγνωρισμού, δηλαδή θα εξετάσει εσείς το θέμα της ε, της, ε, της ε, στάθμισης μεταξύ των Αμερικανικών και των Ευρωπαϊκών ε, δεδομένων. Και το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε για το Standard Poor's γιατί μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας προσπάθησα να υποβάλω κάποιες ιδέες όσον αφορά τους δείκτες και πού θα μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί για καλύτερα, πιο ανοιχτά διεθνή πρότυπα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν καμιά φορά ε, πνευματικά δικαιώματα και γι' αυτό οι άδειε που δεν θα πρέπει να είναι κάπως αναλογικά. Έχουμε κάποια πρότυπα σε αυτό το τομέα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτά είναι ευθυγραμμισμένα με αυτά που έχετε εσείς κατά νου και γενικά όσον αφορά τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα περάσουμε σε ένα σύστημα που θα έχουμε πιο ασφαλή ε, παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικό να έχουμε τα σωστά διεθνή στοιχεία και να τα χρησιμοποιούμε κιόλα. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη ερώτηση. Δεν μπορώ να πω τίποτα για μια προτινόμενη συγχώνευση που δεν μας έχει ακόμα κοινοποιηθεί να πω δύο λόγια για αυτή τη συζήτηση που είναι σημαντική για το επιχειρηματικό μοντέλο, business model για τα, αποθετή, για τα clearing houses κλπ. Από την σκοπιά του ανταγωνισμού προτιμώ μοντέλα τα οποία δεν έχουν κατακόρυφη μορφή γιατί έτσι δημιουργούνται πιο πολλές ευκαιρίες ένα πιο ανοιχτό επιχειρησιακό μοντέλο. Από την πλευρά του ανταγωνισμού είναι προτιμότερο αυτό, η διαλειτουργικότητα του μοντέλου. Από τη συζήτηση βγαίνουν μερικά στοιχεία, παράμετροι που τα συζητάτε και εσείς και στο Συμβούλιο. Π.χ. η αρχική μας πρόταση ήταν σχετικά συνετή για το θέμα αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα και εσείς και στο Συμβούλιο ακούγονται εδώ φωνές που θα το δεχόντουσαν. Αυτό όμως εξαρτάται από τους νομοθέτες που είστε εσείς να αποφασίσετε. Εγώ μπορώ να πω τη γνώμη μου ως αρχή ανταγωνισμού θα προτιμούσα να μην έχω να επιλέξω αυτή την ε, ε, λύση του χαρακτήρα του vertical. Και γι' αυτό ένας λόγος είναι αυτός που επέμενα στην απάντησή μου στον Πίτερ Σκίνερ και σε άλλους ε, ευρωβουλευτές λέγοντας ότι στη διάρκεια της διαδικασίας που θα κάνουμε την ανάλυση πρέπει να έχουμε επαφές με την υποτιθέμενη προσκοινοποίηση συγχώνευση. Δεν είμαι καν σίγουρος αν θα μας το κοινοποιήσουν. Αν μας το κοινοποιήσουν για τη συγχώνευση του χρηματιστηρίου θα το δούμε. Γιατί σίγουρα αν συμβεί αυτό θα είναι πολύ σημαντικό γιατί για τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτής της συγχώνευσης αλλά έχει σημασία και για το μέλλον, για τα για τις δραστηριότητες όσον αφορά την πώληση παραγόγων. Standard and Poor's. Έχω μια συγκεκριμένη περίπτωση. Στο, ε, έχει σχέση με το identification numbers των ε, διεθνών χρεογράφων, επειδή αυτοί έχουν ένα, ένα μονοπόλιο στο να δίνουν αυτούς τους κωδικούς, κατά τη γνώμη μας, χρεώνουν υπερβολικά για τη χρήση αυτών των ε, ταυτοποιητών και οι χρήστες θα πρέπει να πληρώνουν μια συνδρομή αν και δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ έχουμε κατάχρηση. Και το συζητάμε με τους Standard Poor's, αναλύουμε την περίπτωση και δεν αποκλείω να λυθεί το πρόβλημα αυτό με τις Standard Poor's. Δεν αποκλείεται. Από τις επαφές που έχουμε τώρα με τον πρόεδρο αυτής της εταιρείας Μα αναφέρεται και αυτή η πιθανότητα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε τίποτα δεδομένο. Θα σας πληροφορήσω καθοδόν, δεν θέλω να προδικάζω τίποτε. Αν το θέμα των δικτών αυτών, των indexes, απαιτεί άλλου είδους μεταχείριση από τη σκοπιά του ρυθμιστή, τότε αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι δεν είναι μόνη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αυτού του είδους των πινάκων ίντεξης το χρησιμοποιεί είτε για να αποκλείσει ανταγωνιστές ή για να λειτουργήσει με καταχρηστικά στον χώρο της αγοράς. Δεν είναι η μόνη περίπτωση. Πρόεδρος. Βέρνερ. Κύριε Επίτροπε, η ερώτησή μου για την ίση μεταχείριση στον τομέα των τραπεζών δεν χρειάζεται να υποβληθεί γιατί απαντήσατε ήδη. Θα ήθελα να αναφερθώ ένα άλλο τομέα της δραστηριότητά σας όσον αφορά τους όλους τους ανταγωνισμούς της δημόσιας ε, αγοράς. Έχετε την αρμοδιότητα για συγχωνεύσεις, για κρατικές ε, ενισχύσεις και εντάξει και αυτό νομίζω, παρόλο που ίσως ε, προβλέπτουμε στα πλαίσια της ιστορικής αγοράς. Βλέπουμε ότι ιδίω στα νέα κράτη-μέλη έγιναν ε, δημοσίευσεις για δημόσιες αγορές, ιδίως όσον αφορά παραδείγματος χάρη τι υποδομέ ε, μεταφορών στην Πολωνία, στι οποίε οι ευρωπαϊκέ εταιρείε δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν γιατί οι προσφορές ε, υπευλήθησαν εν μέρη με εργαζόμενους από την Κίνα που δεν υπόκεινουν στου ίδιου όρου αναγωνισμού και μισθολογικής ε, ε, εισφορά. Αυτά ε, βέβαια όσον αφορά τον λογισμό είναι πολύ άσχημα. Το ίδιο ισχύει και για ενισχύσει για ε, Έλληνες για την αγορά δυναμικού ως την Νότιο Κορέα πληρώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια. Δεν είναι άμεσα δική σας αρμοδιότητα, έχει όμως σημαντικές επιπτώσεις στον, ε, στο ανταγωνιστικό δυναμικό της ε, ευρωπαϊκής Βιομηχανία. Σας είχα στείλει και σχετικές επιστολές. Επαναλάβατε ότι προτίθεστε να συνεργαστείτε και θα ήθελα να σας παρακαλέσω η Κομισιόν να αντιδρά πιο γλίγορα από ό,τι μέχρι τώρα σε γραπτές και προφορικές επερωτήσεις βουλευτών. Μπορώ να σας πω ότι στην χώρα μου ε, ε, κάτι που έγινε παραδείγματο χάρη ε, δύο βουλευτές υπέβαλα μία επερώτηση για μία για, τα για καταχρηστικές μάλλον κρατικές ενισχύσεις ε, που δόθηκαν σε μια κατασκευή αθλητικού χώρου στο Nürburgring πριν από έξι μήνες και η μόνη απάντηση που ε, πήραμε είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν υπό εξέταση το θέμα. Παρακαλώ να αντιδράτε πιο γλίγορα να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεν. Το πρώτο θέμα που ρωτάτε δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Είναι αρμοδιότητα του Μισελ Μπαρνιέ, που είναι υπεύθυνο για την εσωτερική αγορά. Είναι μια περίπτωση που αναφέρεται πολύ. Και αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο υπάρχει ανησυχία. Ότι τρίτες χώρες μπορεί να επωφεληθούν από το άνοιγμα των δικών μας δημοσίων συμβάσεων, των ρυθμίσεών μας, των προϋποθέσεών μας ενώ σε κάποιες χώρες από όπου προέρχονται επιχειρήσεις που υποφελούνται από τις δικές μας δημόσιες συμβάσεις, δεν υπάρχει τέτοιο άνοιγμα. Και οι δημόσιες συμβάσεις εκεί είναι κλειστές στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και αντιλαμβάνομαι την ανησυχία σας, αλλά και, θα το ξέρετε, αλλά σας το λέω και εγώ, το επαναλαμβάνω, ότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ για την εσωτερική αγορά και ο Κάρελ Τεγκούχτ για το εξωτερικό εμπόριο συνεργάζονται ακριβώς για να λυθεί αυτό το ζήτημα και να βρούνε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από την πλευρά μας να αντιδράσουμε. Τέτοιου είδου αντιδράσεις έχουν δύο δυνατότητες. Η μία είναι να καθορίσουμε μία στρατηγική και να υιοθετήσουμε αποφάσεις προκειμένου να προσπαθήσουμε οι άλλοι να δέχονται τους ανοιχτούς δικούς μας κανόνες και αυτό είναι το θετικό, αυτό το δρόμο πρέπει να πάρουμε. Η άλλη επιλογή που ακούγεται μερικές φορές, αλλά είναι σε βάρος των σιδερόντων μας πιστεύω, είναι να πούμε ότι αφού οι άλλοι δεν τηρούν στις χώρες τους, στις αγορές τους, τους κανόνες που έχουμε εμείς στη δικιά μας εσωτερική αγορά, θα αλλάξουμε τους δικιούς μας κανόνες και θα βάλουμε φραγμούς. Εγώ νομίζω ότι από κάτι τέτοιο πρώτοι από όλους θα πληγούμε εμείς. Νομίζω ότι η σωστή λύση είναι να δουλέψουμε ώστε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο και να από τους εταίρους μας, τους εμπορικούς, τους οικονομικούς, να τηρούν στις δικές τους αγορές τους κανόνες του παιχνιδιού, όπως κάνουμε και εμείς και τους τηρούμε στη δικιά μας εσωτερική αγορά. Και στις δημόσιες συμβάσεις γίνεται. Και γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις όπου έχουμε συζητήσει πολύ, όπου μια κινέζικη εταιρεία η οποία φαινόταν ότι θέτασε σε ανταγωνισμό με δύο ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις για να αγοράσει μια τρίτη στην Ολλανδία. Τελικά δεν μπήκε στον ανταγωνισμό αυτό η κινέζικη εταιρεία, αλλά μπήκε σε συζήτηση το θέμα. Τι κάνει κανείς σε αυτή την περίπτωση. Ε, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από τους άλλους να εφαρμόζουν το ίδιο ανοιχτό πλαίσιο που έχουμε και εμείς στην Ευρώπη. Έχουμε μηχανισμούς σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατεύουμε τα συμφέροντά μας, εθνικά, που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, για να προστατευόμαστε από εξωτερικές επενδύσεις που μας θέτουν σε κίνδυνο, μεν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να ελέγξουμε όπως κάναμε παλιά τις ξένες επενδύσει. γιατί είναι σε βάρος των δικών μας των συμφερόντων. Εμείς επενδύουμε περισσότερο προς τα έξω από ό,τι απ' έξω επενδύουν στην Ευρώπη και έχουμε πολύ περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δουλεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι επιχειρήσεις μη ευρωπαϊκές που δουλεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν προσπαθήσουμε να αντιδράσουμε στα γεγονότα αυτά που είναι ανησυχητικά και χρειάζονται κάποια αντίδραση από την πλευρά μας, αλλά να αντιδράσουμε αμυντικά, πρώτα απ' όλους θα χάσουμε εμείς είναι όπως οι κακές ομάδες στο ποδόσφαιρο που νομίζουν ότι θα κερδίσουν ε, την ε, Μπάρσα ε, παίζοντας αμυντικά. Αν δεν. Τώρα για την περίπτωση του Νομαρίν. Μου έχουν έρθει πολλές επιστολές. Αναλύουμε. Αλλά όταν βλέπετε δεν έχει λυθεί μία περίπτωση ακόμα, είναι πολύ δύσκολο να σας πω πώς θα τελείσουμε. Πολύ θα ήθελα να λύνω σε ένα μήνα τα προβλήματα υπάρχουν περιπτώσεις που λύνονται σε μικρό χρονικό διάστημα και άλλες για διάφορους λόγους, που είναι πιο περίπλοκες περιπτώσεις, αργούν περισσότερο. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Είμαστε κοντά στη λύση σε μία απόφαση. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε και σε κανέναν άλλον πώς θα λυθεί η περίπτωση αυτή γιατί δεν έχουμε φτάσει στη λύση. Αυτά έχω να σας πω. Ο Βάρεν έχει μια συμπραγματική ερώτηση νομίζω. Ναι. Το πρόβλημα κύριε Επίτροπε είναι, αναφερθήκα στον κύριο Μπαγκέ. Ναι, σωστό. Αλλά δεν υπάρχει βέβαια επαρκή συντονισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό και όσον αφορά αυτού του διαγωνισμού και όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει. Δικαίω ασχολείστε με ενισχύσει από κρατικέ υπηρεσίε των κρατών μελών που οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, αλλά το θέμα αυτού του διαγωνισμού στην Πολωνία για 20 δισεκατομμύρια ευρώ που ε, δόθηκε σε μια κινέζικη εταιρεία που οι εργαζόμενοι ε, παίρνουν πραγματικά ψίχουλα χρηματοδοτείται όμως από την Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Για το Nürburgring, την περίπτωση αυτή, το ίδιο σε πιο μικρό ε, ε, σε πιο μικρή κλίμακα. Γιατί ήταν πάλι ένα θέμα των ε, κρατικών ενισχύσεων που αδίκως καταβάλλονται. Εδώ και ένα χρόνο είπε πως υπόσχεση αυτή ένας υπουργός παραιτήθηκε πριν από ένα χρόνο. Έχετε κάνει τίποτα το μεταξύ για να η ειδοποίηση στην γενική κυβέρνηση. Θα επαναλάβω ότι δουλεύω στις υπηρεσίες μου, γιατί είναι δικιά μου δουλειά, για την τραπέζα. Το άλλο όμως της δημόσιας σύμβασης δεν είναι θέμα δικό μου. Η Επιτροπή συντονίζει πολύ καλά τις δραστηριότητε της και γι' αυτό ο κάθε Επίτροπος ασχολείται με τη δικιά του δουλειά και όχι με εκείνη του άλλου. Ο καθένας ξέρει τι κάνουν οι άλλοι, μεν, αλλά δεν κάνει ο καθένας και λίγο από τη δουλειά των άλλων. Το θέμα της κινηζικής προσφοράς με τις πολωνικές αρχές δεν είναι θέμα κρατικής ενίσχυσης, είναι ένα θέμα δημόσιων αγορών, άρα εσωτερική αγορά. Καλημέρα, Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Είπατε κάτι στην αρχική σας παρουσίαση για αεροδρόμια. Είναι ένα θέμα που είναι αρμοδιότητα των χωρών ε, μελών, από όσο ξέρω. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Γιατί όπως ξέρετε στην Ισπανία δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών αεροδρομίων και όπως τα ξέρουν οι συνάδελφοι εδώ, η διαχείρισή τους γίνεται από έναν κεντρικό φορέα. Και αυτά πήγαιναν πολύ καλά μέχρι που ξεκίνησε η κρίση και άρχισαν οι απώλειες. Και τώρα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Και όχι μόνο η Ισπανία, ολόκληρη η Ευρώπη πλήττεται από την έλλειψη ανταγωνισμού. Στην Καταλωνία είναι ευαίσθητο θέμα αυτό πάντως. Και σας ρωτάω, από πλευράς της Ισπανικής κυβέρνησης φαίνεται ότι προτιμάνε να ιδιωτικοποιήσουν το μονοπόλιο αντί να αποκεντρώσουν την διαχείριση και να τη δώσουν στις αυτόνομες περιφέρειες. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, τα Λάντερς διαχειρίζονται σε ένα βαθμό σε ορισμένες περιπτώσεις τα αεροδρόμια. Αυτή θα ήταν μια καλή λύση και θα μας επέτρεπε να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα των αεροδρομίων. Εγώ θα συμφωνούσα με αυτό. Οπότε ρωτάω τον Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό, που είναι και άνθρωπος της αριστεράς, τι πιστεύει. Συμφωνούμε και οι δύο, είμαι βέβαιος. Ο κύριος Λάγκ εκπλήσεται που με είπατε άνθρωπο της αριστεράς. Γιατί γελάτε. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας επίτροπος αριστεράς. Παρεμβάσει εκτός μικροφώνου, δεν τις ακούμε όλες. Λοιπόν, για να απαντήσω στην κύριο Τρεμόσα. Συμφωνούμε σίγουρα και εσείς και εγώ στο εξή. Ό,τι είναι μιας πολιτικής εξουσίας σε χαμηλότερο επίπεδο δεν πρέπει να εξετάσετε από μια εξουσία υψηλότερου βαθμού. Σε αυτό συμφωνούμε, έτσι. Αυτά που με ρωτάτε για τα ισπανικά αεροδρόμια είναι θέμα της Ισπανίας, των ισπανικών αρχών, των κεντρικών, των αυτόνομων περιφερειών ε, κτλ. Δεν είμαι εγώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα το λύσω αυτό. Είναι αποφάσεις που παίρνει ο καθένας στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων, στο δικό του το επίπεδο. Και είμαι πάρα πολύ προσεκτικό, δεν θέλω να παρέμβω και να ανακατευτώ ούτε στις αρμοδιότητες των συναδέρφων μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ούτε στις αρμοδιότητες και τις ευθύνε που εμπίπτουν σε άλλα επίπεδα, στο εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Αυτό όμω που είπα και το επαναλαμβάνω είναι ότι κοιτάω τι γίνεται με τις κρατικές ενισχύσεις στα αεροδρόμια. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ε, περιπτώσεις που είναι ανοιχτέ. Ξέρετε, στην αρχή για τον ανταγωνισμό ασχοληθήκαμε με τις κρατικές ενισχύσεις στις μεταφορές. Από τις κρατικές ενισχύσεις, που έχουμε πολλές, ε, πάρα πολλή δουλειά, υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με αεροδρόμια ή με αεροπορικές γραμμές πολύ φτηνές, χαμηλού κόστους. Και με άλλες κανονικού κόστους, λύθηκαν πολλές περιπτώσεις, αλλά χαμηλού κόστους ιδιαίτερα. Και περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με αεροδρόμια έχουμε πάρει πάρα πολλές. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι μεταξύ άλλων πρέπει να προετοιμαστούμε και να εγκρίνουμε κάποια στιγμή προσανατολισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις που πάνε στα αεροδρόμια. Και για τα λιμάνια επίσης. Δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη θέση. Νομίζω ότι πρέπει όμως, ότι είναι αναγκαίο. Και ξεκινάμε. Τι είναι υποδομή σε ένα αεροδρόμιο και τι δεν είναι. Που μπορούν, που δεν μπορούν να πάνε κρατικές ενισχύσεις. Υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για θέματα ασφάλειας. Στα αεροδρόμια πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι υποδομές, που είναι ο δρόμος ας πούμε που υπάρχει. Εκτός αν υπάρχει βέβαια από κοινού διαχείριση, εντάξει αυτό είναι κάτι άλλο έτσι, τα βλέπει ένα κράτος με τον προπολογισμό του, τι πληρώνει στις περιπτώσεις των αεροδρομίων. Αυτό πάντως που ισχύει είναι ότι υπάρχει και ένα τμήμα που δεν είναι υποδομές και που έχει να κάνει με την αγορά. Και εκεί δεν πρέπει να υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις. Αυτή είναι λοιπόν μία ανάλυση που θα κάνουμε, που είναι πολύ σοβαρή. Ξεκινάμε τις ε, μελέτες, συζητάμε στο τμήμα μου. Δεν νομίζω ότι θα είναι για φέτος, αλλά κάποια στιγμή σίγουρα θα έχουμε πράγματα να πούμε. Θα γίνει και διαβούλευση με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, εννοείται, και θα καταλήξουμε σε κάποιους προσανατολισμούς. Για το 2012 το βλέπω ή και μετά, όχι για φέτος. Αναγνωρίζω όμως και συμφωνώ μαζί σας αυτό, όχι μόνο για το πρώτο, αλλά και γι' αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί πάνε πολλά χρήματα σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Ευχαριστούμε. Κλείνω τον κατάλογο μιλητών τώρα. Έχω την κυρία Κράτσα, και Ζαν Πολ Και νομίζω ότι έτσι θα τηρήσουμε το χρόνο μας. Κύριε Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με συγχωρείτε πολύ αν σας ε, υποβάλω μια ερώτηση με την οποία έχετε ήδη ασχοληθεί, διότι επειδή είχα ψηφοφορίε σε άλλη επιτροπή, ήρθα καθυστερημένη στη συζήτησή σας. Ε, ήθελα να ρωτήσω για το επίκαιρο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Ε, πώς αυτό το σύμφωνο το βλέπετε εσείς, ε, ποια προστιθεμένη αξία μπορεί να έχει σε αυτά που ήδη υπάρχουν ε, σαν πολιτικές στην ε, Ένωση και κυρίως ε, πώς θα ενταχθεί ή θα δώσει παραπάνω στοιχεία από αυτά, τα ήδη, από αυτά που ήδη συζητούμε στο πλαίσιο της, του πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης, στο οποίο, όπως γνωρίζετε, υπάρχει και η πτυχή των, της αντιμετώπισης των ε, ανισορροπιών των οικονομικών πολιτικών, πέρα από τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τι καινούριο εσείς θα περιμένατε από ένα σύμφωνο ανταγωνιστικότητας σήμερα ε, και πώς θα μπορούσε να ενταχθεί αυτά τα καινούργια στοιχεία να ενταχθούν στο πλαίσιο της διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτό που με ρωτάτε Πρέπει να το ρωτήσετε στον Όλυ Ρεν, στο συνάδελφο. Το σύμφωνο που ονομάστηκε Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, ή Σύμφωνο για το Ευρώ, αποτελεί τμήμα αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου για τα οικονομικά ζητήματα. Το 2009 θα σας το απαντούσα εγώ το ερώτημα αυτό. Τώρα όμως το 2011 πρέπει να σας το απαντήσει όλοι Ρεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ ό,τι πει ο Λιρέν και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βρίσκει σύμφωνο. Είναι δικιά του αρμοδιότητα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Πού είναι δικιά σας αρμοδιότητα. Και είναι το λεγόμενο Dowry. Το 80 είδαμε ότι κάθε φορά που το 1980 και μετά πολλές φορές γινόταν ιδιωτικοποίησαμε με επιχειρήσει και παίρνανε επιπλέον ενισχύσεις οι επιχειρήσεις αυτές. Με την λεγόμενη πρικοδότηση που είχαμε εκείνη την εποχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Τα πρόσφατα χρόνια είδαμε και διαπιστώσαμε ελευθέρωση του τομέα. Είχαμε τη Royal Mail ταχυδρομεία στο Βέλγιο, στην Γαλλία με απελευθέρωση εκεί. Πράγμα το οποίο όμως οδήγησε σε δυσκολίες στις συνταξιδοτήσεις. Τέτοια φαινόμενα λοιπόν όπως η περίφημη πρικοδότηση τότε. Πώς επηρεάζει τον οικονομικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι οι κυβερνήσεις απέκτησαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είτε στο σύνολό του έγιναν ιδιοκτήτε τους, είτε σε ένα βαθμό, παίρνοντα μετοχέ. Και μετά ιδιωτικοποιούμε. Οπότε εσείς τι λέτε, ανάμεσα σε αυτή την πυρηνικοδότηση που είχαμε τη δεκαετία του 80 και την εξέλιξη στη συνέχεια με το τι έγινε στα ταχυδρομεία μέχρι το 2011 που φτάσαμε στην ελευθέρωση του τομέα, πιστεύετε ότι κάτι αντίστοιχο θα δούμε και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σαν προειδοποίηση το λέω γιατί εφόσον έγινε η πρικοδότηση νωρίτερα και άμα ξεκινήσει είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε πίσω. Θέλω λοιπόν τη δικιά σας άποψη για το φαινόμενο αυτό και πώς το φαινόμενο αυτό θα το διαχωρίσουμε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Άκουσα στα γαλλικά αυτά που είπατε και δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσατε με τον Τάιρι, λέει ο Επίτροπος. Να σας εξηγήσω τι εννοώ, λέει ο κύριος Έπινγκ. Μπράτσχαρτ στα Ολλανδικά, Ντάουρι στα Αγγλικά και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όταν μια επιχείρηση, το ταχυδρομεία για παράδειγμα, ιδιωτικοποιούνται και από κρατική επιχείρηση γίνεται ιδιωτική επιχείρηση, τότε η κυβέρνηση δίνει κάτι παραπάνω, η πρίκα που είπαμε. Δίνει κάτι παραπάνω σαν ε, βοήθεια είτε πρόκειται για τα γερμανικά ταχυδρομεία, είτε πρόκειται για κάτι άλλο, για να βοηθηθεί και να γίνει πιο δυνατή επιχείρηση αυτή στην ελεύθερη αγορά. Γιατί από κρατική επιχείρηση γίνεται ιδιωτική και πρέπει να είναι εύρωστη. Ένα πουγγί τέλο πάντων της δίνει το κράτος για να μπορέσει να αντέξει στον ανταγωνισμό. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Εντάξει, τώρα που τα άκουσα στα ισπανικά τα κατάλαβα από όλα. Ευχαριστώ πολύ τους Ισπανούς διερμηνείς, λέει ο κύριος Αλμούνια. Πράγματι, αυτό είναι ένα από τα στοιχεία... Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό είναι μια αποζημίωση για έναν ιδιωτικό τομέα που αναλαμβάνει μια κρατική επιχείρηση. Στην περίπτωση λοιπόν ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων που ήταν παλιά κρατικά μονοπόλια και τα οποία έγιναν ιδιωτικές επιχειρήσεις και αναλαμβάνουν μια οικονομική υπηρεσία κοινοφελή, κοιτάμε να δούμε σε τι επίπεδο υπάρχει αυτή η αποζημίωση, η αντιστάθμιση. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις. έχουμε αναλύσει πολλές περιπτώσεις, σαν και αυτές τις οποίες αναφερθήκατε. Οι συνταξιούχοι που περνάνε από ένα σύστημα σε ένα άλλο, μερικές φορές αυτό έγινε με κάποιες επιδοτήσεις προς έναν φορέα, που είναι ένας ιδιωτικός φορέας βέβαια, Άλλες περιπτώσεις, άλλα σενάρια που είδαμε, είναι ότι αυτές οι υπεραντισταθμίσεις γίνανε διασταυρωτά. Δηλαδή στην αρχή ήταν η κοινοφιλής υπηρεσία που έπαιρνε μια επιδότηση, αλλά τελικά η επένδυση έγινε για να μπορέσει η συγκεκριμένη επιχείρηση όταν βρεθεί στον ανταγωνισμό σε άλλους τομείς να αντέξει. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις τέτοιες που έχουμε λύσει και άλλες που εξακολουθούμε να αναλύουμε. Τα ταχυδρομεία, για παράδειγμα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές περιπτώσεις. Τα βέλγικα ταχυδρομεία και τα γερμανικά ταχυδρομεία. Είναι δύο παραδείγματα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Θα μπορούσα να σας αναφέρω πολλά άλλα παραδείγματα και σε άλλους τομείς. Είναι πάντως πολύ σημαντικά. Πάντως, στην αρχική μου παρέμβαση, όταν είπα ότι το σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε στους μεγάλους φορείς. Αυτό εννοούσα, βασικά τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ενώ δεν έχει και πολύ σημασία να δίνει κανείς ε, χρόνο ενέργεια για να εξετάσει μια μικρή επιχείρηση που δρά τοπικά και προσφέρει τοπικά υπηρεσίες και παίρνει κάποια επιδότηση από το Δήμο. Από το Δήμο της. Κάτι τέτοιο δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, δεν επηρεάζει τις συναλλαγές μέσα στην εσωτερική αγορά. Οι πολίτες στο συγκεκριμένο Δήμο θα φροντίσουν οι δήμαρχοί τους και οι δημοτικοί του σύμβουλοι να διαχειρίζονται σωστά τα χρήματα. Για να χρησιμοποιείτε καλά το δημόσιο χρήμα, πρέπει να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας σε τέτοιες περιπτώσεις ε, άρρητων ε, επιδοτήσεων. Κρυφών, που μερικές φορές κατέληξαν σε στρεβλώσεις και σε αρνητικές συνέπειες. Τέτοιοι μεγάλοι φορείς κοινοφελών υπηρεσιών πρέπει να τραβήξουν την προσοχή μας, γιατί είναι κάτι που δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική ροή, αλλά έχει να κάνει και με την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε ένα επίπεδο επιδοτήσεων για ένα συγκεκριμένο βαθμό αποτελεσματικότητας, αλλά αν η αποτελεσματικότητα, η απόδοση του τομέα δεν είναι καλή, δεν βλέπω γιατί να κρατάμε το ίδιο επίπεδο ε, δημόσιας ε, επιχορήγησης. Είναι θέματα αυτά τα οποία μας απασχολούν και μας προβληματίζουν. Ευχαριστούμε ο Ζαν Πολ Ευχαριστώ κύριε Πίτρεπε που απαντήσατε. Σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή και γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα σας. Ακούγοντας όμως κόβουμε στα δύο μέσα μου και σκέφτομαι τον πολίτη που συναντάμε συχνά γιατί αντίθετα με αυτά που λένε πολλοί οι ευρωβουλευτέ συναντάνε του πολίτε και μιλάνε με αυτού, υπάρχει το δικαίωμα ανταγωνισμού για τις ελίτ και υπάρχει το πώ το αντιλαμβάνεται τον ανταγωνισμό ο πολίτη, ο μικροεπιχειρηματία. Τα είπε ο Βέρνερ Λάγκεν πιο πριν τα σχετικά. Και πώ αντιλαμβάνεται κανεί την Ευρώπη σήμερα. Ξέρετε, η εικόνα της Ευρώπης είναι κακή αυτή τη στιγμή. Δέτε τα αποτελέσματα των εκλογών στι διάφορε χώρε. Και λέω, θα πρέπει να έχουμε μια λογικό ανταγωνισμό, όπως μιλάμε για μια λογική γεωργία. Και όπως είπατε πριν, αν υπάρχουν εμπόδια, πάμε χαμένοι. Εδώ μας ζητάτε κάτι να το δεχτούμε τυφλά, ενώ οι πολίτες τι βλέπουνε. Χάρη στο άνοιγμα της Ευρώπης, που είναι σημαντικό, δεν μπορούν να αντιληφθούν όλα τα ωφέλη. Δεν υπάρχει αναγκαία αμοιβαιότητα. Δεν λέω να αμφισβητηθεί ο ανταγωνισμός. Αλλά λέω εκεί που είμαστε σήμερα, με τις δυσκολίες που ζούμε, σε όλες τις χώρες μας, οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν τι νόημα και τι χρησιμότητα έχει ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη. Δεν σα κατηγορώ, αλλά θυμάμαι στην προηγούμενη εντολή σα, το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο για τον ανταγωνισμό στην Επιτροπή, συχνά στι συνεδριάσει άρχιζε και σε ευχαριστώ που δεν το κάνετε λέγοντα, αυτό το τρίμηνο κατάφερα να επιβάλλω τόσα εκατομμύρια πρόστιμα. Και μία φορά τόλμησα να ρωτήσω, ο καταναλωτής κέρδισε τίποτα από την ιστορία αυτή. Και από ό,τι θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος, να μην θυμάμαι καλά, μου απάντησε ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι πολιτική εφαρμόζει σήμερα η Ευρώπη και αν η πολιτική για τον ανταγωνισμό που ασχεί την καταλαβαίνει ο πολίτης και αν ωφελείται και αν βοηθάει τον οικονομικό ιστό. Γιατί υπάρχουν μεν θεωρητικά επιχειρήματα, αλλά στην πράξη ο κόσμο σε αυτά δεν τα καταλαβαίνει. Περισσότερο σχόλιο αυτό παρά ερώτηση, κύριε Επίτροπε. Επειδή η σχέση μα είναι ειλικρινή και επειδή δουλεύετε σωστά και καλά, έκρινα σκόπιμο να σας το καταθέσω το σχόλιο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Γκοζές. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας απαντήσω πολιτικά, όχι τεχνοκρατικά. Ο ανταγωνισμός για ποιον, υπέρ τίνος του καταναλωτή και του πολίτη και ένας άλλος δικαιούχος, η μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν το λέω κάθε φορά που έρχομαι τα πρόστιμα αλλά πέρυσι το 2010, πρώτο χρόνο εντολής μου ως Επιτρόπος, τρία δις πρόστιμα. Δεύτερη χρονιά υπέχαμε τόσο μεγάλα πρόστιμα. Σε τι τα πρόστιμα. εναντίον αεροπορικών εταιριών που έχουν ένα υπερβολικό κόστος που έβλαψε πάρα πολλές επιχειρήσεις που χρειάζονται τις αερομεταφορές για να εξάγουν και έβαλαν ένα επίναυλο. Οι πολίτες υποφέρουν φυσικά γιατί πληρώνουν πιο ακριβά τελικά οι πολίτες. Την τιμή του εμπορεύματος στο οποίο επιβλήθηκαν ψηλότερες τιμές από ένα καρτέλ εταιρεών που προσπαθούν να ελέγξουν τις αερομεταφορές. Υπάρχουν και άλλες αποφάσεις χωρίς πρόστιμα. Απόφαση για τη συγχώνευση του κλάδου άρθρου ε, ε, φροντίδες για το, για το σώμα, σαμπού και λοιπά, σαμπουάν και τέτοια. Πράγματα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα δηλαδή, τέτοιου είδους φροντίδες σώματος. Και είπαμε δύο μεγάλες εταιρείες. Είπαμε αν θέλετε να δεχτούμε αυτή τη συγχώνευση, θα πρέπει να διαχωρίζετε αυτό τον κλάδο από τον άλλον. Διαφορετικά, η τιμή που θα πληρώνει ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ για τα προϊόντα θα ανέβει. Διότι μέσω αυτής της συγχώνευσης, όπως μας την προτείνετε θα ανέβουν οι τιμές σε πολλές χώρες της Ένωσης. Πολίτες είναι αυτοί, κύριε Γκονζές και οι ευρωβουλευτές, ο επίτροπο και ελπίζω και οι Υπουργοί πρέπει να τα εξηγούν όλα αυτά στον πολίτη. Γιατί ο πολίτης την οικονομία του ανταγωνισμού τις αποφάσεις τη Κομισιόν δεν τα, δεν τα βλέπει, δεν τα μπορεί να τα εξηγήσει μόνο του. Εμεί θα πρέπει να τα εξηγήσουμε και αν του εξηγήσουμε δεν είναι χαζοί, θα το καταλάβουν. Είναι πολύ έξυπνοι οι πολίτε και μερικέ φορέ πολύ πιο έξυπνοι από εμά. Γιατί έχουν την διέστηση ότι είναι προς όφελός τους. Μια μέρα είχα μια συνεδρίαση με πολίτες. Εν πάση πτώση, κάθε φορά που, που συζητάμε, ε, δεν ακούω να διαμαρτύρονται για τα πρόστιμα ή γιατί κινούμαστε κατά τον καρτέλ. Δεν λένε τι κάνετε εσείς εκεί για τον ανταγωνισμό, όχι. Μόνο όταν έχουμε συνεδριάσει με μεγάλε επιχείρησει, εκεί είναι το θέμα. Α, τι κάνει η Ευρώπη για τι συγχωνεύσει, τι κάνει η Ευρώπη με τα πρόστιμα, εκεί αναφέρονται αυτά. Εγώ όμως δεν είμαι ε, ε, επίτροπος που εκπροσωπώ τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είμαι για να προασπίζω τα γενικά συμφέροντα της Ευρώπης, δηλαδή των πολιτών και των δισεκατομμυρίων μικρών επιχειρήσεων που υποφέρουν από την έλλειψη ανταγωνισμού. Το θέμα Ευρώπη, πώς βλέπει ο πολίτης την Ευρώπη. Κάθε φορά που η Ευρώπη δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση, αυτό δεν αρέσει τον πολίτη κάθε φορά που το ΕΚΟΦΗΝ, που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει και στο τέλος δεν υπάρχει απόφαση για να λυθεί ένα πρόβλημα των Ελλήνων, των Ιρλανδών, των Πορτογάλων ή των Λετωνών ή των Ρουμάνων, υποφέρει ο πολίτης και λέει τι κάνει η Ευρώπη. Αν και ελπίζω να συμβεί αυτό, αν τις επόμενες μέρες οι πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για να απαντήσουν στο, σε αυτά που υποφέρει ο λιβικός λαός. Αν υπάρξει σύγκρουση στο ιστορικό της Ευρώπης, οι πολίτες σωστά θα πούνε τι κάνει η Ευρώπη και εμείς θα πρέπει να πούμε η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη, να αναλάβει τις ευθύνε της, να πάρει αποφάσεις. Κάθε φορά που παίρνει αποφάσεις η Ευρώπη, οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα πρέπει να φύγει προς τους πολίτες και όχι ένα μήνυμα φόβου, ή αμυντικά επιχειρήματα. Γιατί παίζοντα το αμυντικά η Ευρώπη δεν πρόκειται να προχωρήσει. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ και έτσι τελειώσαμε με την σημερινή ακρόαση. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που δώσατε. Θα σας ξαναδούμε σύντομα. 12 Ιουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. And we'll have about a five minute διάλειμμα πέντε λεπτών πριν περάσουμε στην ακρόαση Okay, everybody. Λοιπόν, παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Περνάμε στο σημείο 7 της διάταξης που είναι μια δημόσια κρόση για τα στήματα εγγύησης των καταθέσεων, συμβολή στην γραμματοπιστωτική σταθερότητα, διασφάλιση εμπιστοσύνη των καθαθετών. Με μεγάλη ευχαριστήση θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τους εμπειρογνώμονες. Ο Ντερ Κουπέ που είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Βήματος Ασφαλιστών Αποταμιεύσεων που θα μας κάνει μια εισαγωγή 15 λεπτών. Μετά θα προχωρήσουμε να ακούσουμε την Βέρα Κοτσουέλ 10 λεπτά να μας παρουσιάσει την ε, πολιτική της WITCH για να ε, εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των ιδιωτικών αποτεμφιών και μετά θα έχουμε ένα πάνελ σε δύο τμήματα, καταρχήν ο Αντρέας Πάγκαλ και ο Φεντερίκο Κορνέλη που θα μιλήσουν για τη δημιουργία μιας, ενός σχεδίου θεσμικής προστασίας για τις Ιταλικές ε, Συνδριστικές Τράπεζες και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα, Λουίς Τεβέγκα, από σκοπιά της ε, τραπεζικής, ε, της ισπανικής συγγνώμη, τραπεζικής αγοράς και μετά έρωτα ερωταποκρίσεις. Πολύ πυκνό πρόγραμμα λοιπόν, παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σας. Πρώτος μιλήσει 15 λεπτά και οι άλλοι 10 λεπτά. Και μη διαβάζετε παρακαλώ το έγγραφο σας τόσο γλίγορα που δεν θα προφτάσουν οι διερμηνείς να σας ε, παρακολουθούν γιατί θα αναγκαστώ να σας διακόψω. Χωρίς να σας δώσω περισσότερο χρόνο κόρευσης. Λοιπόν, όταν με βλέπετε να απελπίζομαι, παρακαλώ να ολοκληρώσετε την παρουσία σας γιατί θα πρέπει να έχουμε και χρόνο για αποκρίσεις. Χωρίς περισσότερη εισαγωγή θα ήθελα να περάσω στον πρώτο εισαγωγή αγορητή, τον Dirk Κουπέιν. Λυπούμε, ίσως δεν έχω προφέρει σωστά τα ονόματά σας, αλλά τι να κάνουμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια παρουσίαση για την πρόταση της έκθεσης και το θέμα της εγγύησης των αποταμιεύσεων. Καταρχήν θέλω να πω σας δύο στο για το ευρωπαϊκό βήμα, αυτό το έφτι που ίσως δεν γνωρίζετε, European Forum Deposit Insurers, Ευρωπαϊκό Βήμα Ασφαλιστών Αποταμιεύσεων εκπροσωπούνται όλοι εκείνοι που ε, ασφαλίζουν και εγγυούν από τα μειωτικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 57 συστήματα από 52 χώρες, εκ των οποίων 40 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΦΤΗ ιδρύθηκε το 2002, εργάζεται πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έργο μας είναι ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και εξασφάλιση των ε, τα συστημάτων εγγύησης στην Ευρώπη σε συνεργασία με τα νομοθετικά όργανα και τους αρμόδιους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΕΦΤ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΦΤ προετοιμάζει και κάποια έγγραφα βασικών θεμάτων παραδείγματο χάρη ενό ανάλογα τον κίνδυνο και τα ασφάλιστρα, διαφοροποίηση των αποτεμίευσεων, συνεργασία μεταξύ των συστημάτων εγγύησης, το θέμα της λεγόμενη public awareness, της γνώσης δηλαδή από το κοινό και διάφορα άλλα σημαντικά θέματα. Τα σχέδια αυτά της FD δεν είναι μόνο καθαρά λεγόμενα pay box, δηλαδή για αμυγή εκταμίευση, αλλά η εντολή μας είναι πολύ ευρύτερη. Ένα μεγάλο τμήμα των συστημάτων εγγύησης έχουν διαφορετικό πλαίσιο. Έχουμε επόπτες των τραπεζών, έχουμε την διαχείριση του χρέους, δημόσια διαχείριση του χρέους που είναι τμήμα των εγγύσεων και έχουμε επίσης ενώσεις των τραπεζών και επίσης ιδιωτικές ε, μονάδες που εγγυούνται επίσης αποταμιεύσει. Είναι τμήμα τουλάχιστον του συστήματος εγγύησης των αποταμιεύσεων. Ε, γι' αυτό σας το λέω για να ξέρω δεν είναι μόνο θέμα τραπεζών, είναι πολύ πιο ευρύ ο τομέα δηλαδή κεντρικές τράπεζες, εποπτικά σώματα, ε, διαχείριση χρεών και ορισμένες, όπως σας είπα, ιδιωτικές επιχειρήσεις. το έργο το ε, εγγύηση από μία στην Ευρώπη είναι διαφοροποιημένο. Το λιγότερο είναι το, λιγότερο, το λεγόμενο paybox για την αμυγή ταμείας δηλαδή. Ε, πρέπει επίσης να παρέμβουν και να υιοθετούν κάποια μέτρα για να μην καταλήξει ε, η, η, η μονάδα αποταμίευσης σε πτώχευση. Επίσης ελέγχουν και εποπτεύουν τα διάφορα αυτά Ινστιτούτα, κάνουν κάποια αξιολόγηση, rating, αξιολογούν το κίνδυνο και ούτω καθεξής. Αυτά όσον αφορά γενικά για την FT. Τώρα θα αναφερθώ στην οδηγία για την εγγύηση των αποταμιεύσεων του 1994. Η οδηγία αυτή ήταν ένα, ε, μια ελάχιστη αναμόνιση των αποταμιεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ορισμένα πράγματα που είναι ελάχιστη προστασία 20.000 ευρώ, ε, νομικό δικαίωμα των ε, αποταμιευτών αλλά ήταν πολύ ευέλικτα, θα μπορούσε δηλαδή να υπήρχε και υψηλότερο επίπεδο προστασίας, πράγμα που έκαναν διάφορα κράτη μέλα, μέλη. Η, η, η δυνατότητα ίδια συμμετοχής, δηλαδή ο ε, πελάτης θα μπορούσε να έχει ο ίδιος μια απώλεια μέχρι το 10% μέσα στα πλαίσια των 20.000 ευρώ και επίσης και η δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης προστασίας όχι μόνο των αποταμιευτών, αλλά και ασφαλιστικών εταιριών, ορισμένων χρηματοπιστικών εντερμάτων κλπ. Εκεί υπήρχε ευελιξία, δηλαδή ορισμένοι από τους κανόνες της οδηγίας του 1994 ήταν υποχρεωτικοί, ορισμένοι ήταν ε, μη υποχρεωτικοί και ευέλικτοι και υπήρχαν και ορισμένα θέματα που έμειναν ανοιχτά, παραδείγματο τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών αυτών συστημάτων, τη εντολή των συστημάτων αυτών, πόσα συστήματα θα πρέπει να υπάρχουν κράτο, ποιο θα είναι ο φορέα εκάστοτε και κατά πόσον θα ήταν δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου τα συστήματα της εγγύησης. Τον Ιούλιο του 2010 υπήρξε μια πρόταση της Κομισιόν για μια οδηγία για την εγγύηση της αμοτομίευσης που προέβλεπε περαιτέρω εναρμόνιση ε, των εγγύησεων αυτών στην Ευρώπη. Ορισμένα πράγματα που δεν είχαν διακανονιστεί εντάσσονται στην οδηγία αυτή, παραδείγματος χάρη το θέμα χρηματοδότησης και ορισμένα άλλα πιο δεσμευτικά και πιο εις βάθος ε, διακανονίζονται όσον αφορά αυτή την πρόταση του Ιουλίου 2010, το κεντρικό θέμα ήταν ότι υπήρχε ένα στόχος 1,5% των λεγόμενων eligible deposits, των δικαιωμένων δηλαδή δικαιούχων ε, αποταμιεύσεων, 150 εκατομμύρια σε 10 χρόνια προβλέπεται μέχρι τότε 18,5 δις υπήρχαν αντί 150 δις που ζητάει τώρα η οδηγία. Ε, προβλέπονται εκτός από τα 18,5 εκατομμύρια συμπληρωματική προσθήκη 5 δισεκατομμυρίων στα συστήματα αυτά εγγύησης. Η Κομισιόν προτείνει ένα σύστημα αμοιβαίας αλληλεγγύης, mutual solidarity, όταν υπάρχει δηλαδή υπάρχει ενό συστήματο εγγύηση, θα πρέπει να υποστηρίζεται από κάποιο άλλο που θα του δίνει μια πίστοση, ένα δάνειο. Το θέμα της αρχής της ε, πατρίδας, όπως λέγεται, αμφισβητείται τώρα, θα πρέπει να υπάρχει ε, αρμοδιότητα και της χώρας υποδοχής όταν υπάρχουν θηγατρικές ε, εταιρείες. Η προθεσμία αποζημίωσης μειώθηκε στις 7 μέρες, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, που σε μεγάλο ποσοστό χαιρετίστηκε από την ΕΦΤΗ, ιδίως όσον το θέμα της εναρμόνισης, όσον αφορά το ύψος της ε, προστασίας των 100.000 ευρώ, το θέμα της υποχρέωσης ε, κοινοποίησης, όλα αυτά έτυχαν θετικές υποδοχές από την ΕΦΤΗ. Αυτό που επικρίνει η ΕΦΤΗ είναι ο ορισμός των καταθέσεων, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ στενός ο ορισμός αυτός, δεν καλύπτει όλα τα ε, χρηματοπιστωτικά προϊόντα που πιστεύουμε θα έπρεπε να καλυφθούν. Επίσης επέκρινε η ΕΦΤΗ το ότι λαμβάνεται σαν βάση το λεγόμενο δικαιούχο, δικαιούχος αποταμίευση, eligible δηλαδή. Επίσης επικρίνουμε την προθεσμία ε, αποζημίωση σε 7 μέρες που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξο γιατί αρχές του 2011 εισήχθη μια υποχρεωτική προθεσμία 20 ε, ημερών και ήταν αδύνατο να μειωθεί τόσο γλίγορα σε 7 μέρες. Υπήρχε και υπάρχει μια βούληση της ΕΦΤΗ να μειωθεί αυτή η περίοδος ε, για την αποζημίωση, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει καταρχήν να εισαγάγουμε το λεγόμενο single customer view, την άποψη του ε, ενιαίου πελάτη, αλλιώς δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν αυτές οι πολύ στενές προθεσμίες. Επικρίθη επίσης το ύψος ε, της χρηματοδότησης, αυτό το 1,5% δηλαδή, και επίσης το ύψος της ενδεχόμενης υποχρέωσης ε, συμπληρωματικής καταβολής κατ' έτος, το σύστημα των υποχρεωτικών ασφαλίστων, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει υπερβολική, υπερβολικός από το κράτος πιστεύουμε ότι τα συστήματα υγείας θα πρέπει να προσαρμοστούν διαφορετικά. Επίσης, ε, επικρίθηκε το θέμα της λεγόμενης αμοιβαίας αλληλεγγύης. Επικρίθη από την ΕΦΤΗ πολύ έντονα η υποχρέωση ε, του τρόπου μάλλον επενδύσεων των ποσών αυτών εγγύησης, γιατί ποτέ στην Ευρώπη δεν υπήρχε επένδυση των ε, ασφαλείς των που οδήγησαν σε απώλειες και γι' αυτό δεν θεωρεί αυτή ότι χρειάζεται τώρα να υπάρχουν τόσο ευρύς ε, κανόνες. Επικρίθηκε επίσης από την ΕΕ το θέμα της αρμοδιότητας της χώρας υποδοχής, της δεσμευτικής αρμοδιότητας της χώρας ε, υποδοχής συμπνόχευση θηγατρικών εταιριών Υπάρχει κάποιο σχέδιο της συνεργασίας ε, των ε, εγγυητικών οργανισμών και πιστεύουμε ότι θεωρητικά μπορεί να βρεθεί κάποια δυνατότητα συμμετοχή στι χώρε υποδοχή, αλλά όχι υποχρεωτικά. Επικρίθη από την ΕΦΤΗ επίση ε, το γεγονό ότι θα πρέπει οι πληρωμέ τη αποζημίωση να γίνονται σε όλα τα νομίσματα, όχι μόνο δηλαδή στη χώρα, της χώρας υποδοχής ή σε ευρώ. Αυτό καθυστερεί ακόμα περισσότερο της ε, καταβολής της και επίσης ο περιορισμός των εντολών της, ε, του σώματος εγγύησης με τον περιοριστικό χαρακτήρα της χρήσης των πόρων. Δηλαδή, μέχρι τώρα που να κάτω τέτοιο μόνο αν είχε φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο το ύψος των καταθέσεων. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποια είναι η καλύτερη πρακτική διεθνώς δεν υπήρξε μέχρι τώρα ποτέ περιορισμός ε, των πόρων αυτών ακόμα και η Επιτροπή Βασιλείας ε, που συνεργάζεται για να προετοιμάσει τις βασικές αρχές στην εγγύηση των αποταμνεύσεων που δεν γνωρίζει αυτή τη μέθοδο και ούτε θέλει να την συμπεριλάβει. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να σας πω ότι η ΕΦΤΗ χαιρετίζει έντονα την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί λίγο πολύ όλα τα σημεία επίκρισης του ΕΦΤΗ για την οδηγία αυτή έχουν ληφθεί υπόψη από τον εισηγητή. Ο εισηγητή γενικά ως βάση υπολογισμού όπως συζητήθηκε και στο Συμβούλιο δεν ε, βασίζεται στα λεγόμενα eligible deposits αλλά τα covered ε, deposit. Και αυτό είναι σωστό γιατί μόνο αυτά, τα, αυτές οι καλυμμένες ε, καταθέσεις επιτρέπουν σύγκριση από μία χώρα στην άλλη. Ο εισηγητής προβλέπει επίσης μία ευελιξία που δεν υπήρχε στην πρόταση Κομισιόν κάτω από συγκεκριμένε ε, προποθέσει που ορίζονται και είναι λογικέ. Υπάρχει απόλυτα ελεύθερη χρήση των πόρων. Και κάτι επίσης που βλέπει με κριτικό μάτι η ΕΦΤΗ είναι ότι θα μπορούν τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν και για άλλους στόχους. Χαιρόμαστε που με την πρόταση αυτής της έκθεσης είναι δυνατή η χρήση των πόρων αυτών όπως γινόταν μέχρι τώρα στα κράτη-μέλη και όπως είναι και μία από τι βέλτιστες πρακτικές ε, τη Επιτροπή Βασιλείας. Χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι ο εισηγητής συμπεριλαμβάνει και άλλες λεπτομέρειες ε, στην εκθεσή του παραδείγματος χάρη ότι ε, οι αποζημιώσεις θα πληρώνονται μόνο σε ευρώ ή σε νομίσματα κρατών μελών ότι είναι δυνατή ελεύθερη επένδυση των μέσων σε ρευστό, ότι ιδίως όσον αφορά την συμβουλή για τον ε, κίνδυνο θα χρησιμοποιηθούν τα συστήματα που έχουν αποδειχθεί θετικά στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very um, Ευχαριστούμε πολύ. Οι ερωτήσεις μένουν για το τέλος, για τις 12, έτσι. Να το ξέρετε. Ναι, Βίκυ, έχω δει ότι θες να ρωτήσεις κάτι, αλλά είναι για αργότερα. Συνεχίζουμε και περνάμε στην κυρία Κοτρέλ, που είναι από το WITCH. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να έρθω εδώ σήμερα. Ονομάζομαι Βέρα Κοτσέλ και είμαι σύμβουλος πολιτικής για θέματα οικονομικά στο WICS, που είναι μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση καταναλωτών. Η ευρύτερη είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι πολύ μεγάλη στην Ευρώπη. Είμαστε ανεξάρτητοι από κυβέρνηση, από τον κλάδο και η χρηματοδότησή μας γίνεται μέσω περιοδικών και βιβλίων που πουλάμε για τους καταναλωτές. Είμαι υπεύθυνη λοιπόν για το θέμα αυτό, για τα συστήματα εγγύσεων καταθέσεων στο WITCH. Αποτελεί έναν από τους ακρογωνίους λίθους τρέχουσα, στο τρέχουσα, τρέχον τραπεζικό μοντέλο στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο Αυτά που έγιναν με την Northern Rock το 2007 υπογραμμίζουν πόσο μεγάλη σημασία έχει η εγγύηση καταθέσεων και επίση θέτει και το ερώτημα το τρέχον σύστημα είναι κατάλληλο και πετυχαίνει αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Στην έκθεση αυτή ο εισηγητή προτείνει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση ε, μιλώντας για κοινέ προϋποθέσεις που θα εφαρμόζονται σε όλα τα συστήματα εγγύσεων καταθέσεων, αλλά συγχρόνως θα υπάρχει και ελαστικότητα για να, λειτουργεί, να λειτουργούν τα συστήματα αυτά που θα βασίζεται στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα θα σας μιλήσω για ορισμένα σημεία τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα τους καταναλωτές. Η ελαστικότητα είναι σωστή λύση κατά τη γνώμη μας. Συγχρόνως όμως πρέπει να πω ότι συμφωνούμε και με πολλά από αυτά που λέει ο συγητής, ιδιαίτερα για το θέμα των ε, προπολογισμών, μάλλον των ισολογισμών που είναι προσωρινά υψηλή. Πρέπει να δούμε λοιπόν σε τι επίπεδο επίση πρέπει να γίνεται η παρέμβαση σε περιόδους κρίσης. Θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν στις ε, αρχές του συστήματος εγγύσεων καταθέσεων και πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτές αποτελεσματικά. Οι αγορές έχουν σαν προϋπόθεση την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αυτή η αρχή πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογείται κατά πόσο η αρχιτεκτονική, διαδικασία και τα συστήματα που έχουν να κάνουν με τι εγγύσει καταθέσεων ε, εμπνέουν εμπιστοσύνη στον καταναλωτή ή όχι. Χρειάζεται να υπάρχει ένα προστατευτικό δίκτυο και το οποίο επίσης δεν θα φορτώνει υπερβολικά τον καταναλωτή. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση όσον αφορά τα συστήματα αυτά, αλλά να μην χρειάζεται επιπλέον να κάνει ερμηνεία τους ο καταναλωτής. Ούτε πρέπει να περιμένουμε ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να λειτουργούν με εξουσιοδότηση ή ότι θα αποτελούν οι ίδιοι οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Όχι, θα πρέπει όλοι αυτοί οι φορείς να ξέρουμε ότι δεν έχουν μπορέσει να υπολογίσουν μέχρι τώρα κατάλληλα τον κίνδυνο. Οι καταναλωτές λοιπόν δεν μπορούν να έχουν τη δέουσα επιμέλεια για να εξετάσουν την κατάσταση, άρα δεν μπορούν να ξέρουν ποιος είναι ο κίνδυνος ενός προϊόντος εφόσον αυτός δεν επισυνάπτεται με το προϊόν. Οι καταναλωτές επιλέγουν ε, τα διάφορα τις καταθέσεις που θα δώσουν τα χρήματά τους δηλαδή και που θα κάνουν τις αποτεμιεύσεις τους ανάλογα με τα αποτελέσματα στην επένδυση ενός προϊόντος, αν τα τελευταία 10 χρόνια για παράδειγμα υπήρχε ασφάλεια στην αγορά ή όχι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους καταναλωτές να έχουν τη δέουσα επιμέλεια για να γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση ε, ενός ε, αποταμιευτικού οργανισμού. Θα αναφερθώ τώρα στο θέμα της πληροφόρησης. Υπάρχει στο Μένο Βασίλειο μεγάλη σύγχυση ανάμεσα στον πορικό Σύμβημα μιας τράπεζας και τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών η Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών έκανε μια έρευνα και κατέληξε στο ότι όσοι απάντησαν στην έρευνα αυτή λένε ότι η διάκριση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα υπάρχει χωριστή επεξεργασία της ε, κάθε περίπτωσης. Αλλά εκπλήσονται οι καταναλωτές όταν βλέπουν ότι αυτό είναι δυνητικό και ότι δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει τέτοια διάκριση, πράγμα το οποίο ε, σημαίνει ότι θα υπάρχει μπέρδεμα και δυσκολία στην αποζημίωσή τους. Το θεωρούν άδικο και στη χειρότερη περίπτωση μια πρακτική από την οποία επιφελούνται οι τράπεζε σε βάρο των καταναλωτών. Όσοι απάντησαν στην έρευνα επίση λένε ότι ε, η διάκριση αυτή που γίνεται έχει σαν ε, αποτέλεσμα να καταγγέλουν ε, το γεγονός ότι δεν θα είναι σίγουροι για την αποσημείωση τους οι καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν οι καταναλωτές γιατί λειτουργεί έτσι το σύστημα. Είναι πολύ δύσκολο. Διακόπτη πρόεδρος, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά παρακαλώ γιατί οι διερμηνείς δυσκολεύονται με αυτή την ταχύτητα ενός γραπτού κειμένου. Είναι πολύ δύσκολο, συνεχίζω μιλήτρια, οι καταναλωτές ε, να ξέρουν ποιοι και ποιοι όχι έχουν έναν, την αδειοδότηση, πως παίρνουν την αδειοδότηση διάφοροι οργανισμοί και τι γίνεται με τις ε, συγχωνεύσεις επίσης ε, τέτοιων οργανισμών. Επίσης, από την έρευνα φάνηκε ότι οι καταναλωτές πιστεύουν ότι αν αλλάξει ότι πρέπει να αλλάξει μάλλον η αδειοδότηση, ώστε η κάθε επιχείρηση να είναι εξίσου υπεύθυνη και χωριστά υπεύθυνη για να αποζημιώσει τους καταναλωτές. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι η προστασία πρέπει να είναι στο επίπεδο του καταναλωτή. Η βάσει της κάθε επιχείρησης, του κάθε σήματος, όταν αλλάζουν οι τίτλοι, η ιδιοκτησία, η κατανομή με ένα τρίτο μέρος, τότε το μόνο που γίνεται είναι ότι μειώνεται η προστασία του καταναλωτή και τη συγχυση σύγχυση όσον αφορά αυτήν. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι ορισμένα κράτη-μέλη ζητάνε από τι επιχειρήσει να έχουν χωριστέ άδειε για του διαφορετικού κλάδου του και γι' αυτό προσφέρουν στου καταναλωτέ χωριστά αποζημιώσει. Πιστεύουμε ότι η απουσία μια ε, πανευρωπαϊκή απέτηση να υπάρχουν χωριστέ άδειε για διαφορετικού κλάδου οι ελάχιστε απαιτήσει για κατάλληλη προστασία του καταναλωτή σε όλα τα κράτη-μέλη σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να επιτρέπουν πληρωμέ ανακλάδο και ανακαταναλωτή. Κάτι άλλο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι οι υψηλοί ισολογισμοί προσωρινά. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει κάλυψη και για την περίπτωση αυτή προσωρινά υψηλών ισολογισμών, μια που υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές έχουν ε, σε τέτοιες ε, τράπεζες τις αποταμιεύσεις τους. Ε, θύματα ε, κάποιας εγκληματικής ενέργειας ή μετά από ένα τύχημα ή μετά από μία αποζημίωση ή πληρωμές ασφαλιστικές. Αλλάζει ο ισολογισμός πολύ εύκολα. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά όργανα όπου η προστασία αυτή είναι αναγκαία. Όχι απλώς αιτιολογείται, αλλά είναι αναγκαία για την προστασία των καταναλωτών. Και έτσι χαιρόμαστε που κάνει ε, προτάσεις ο συγκητής στο κείμενό του, όπου λαμβάνει υπόψη και ζητάει μάλλον τον σαφή ορισμό των ε, κατ' ε, προσωρινά υψηλών ισολογισμών και τις προτάσεις της Επιτροπής τώρα. Η πρόταση της Επιτροπής ζητάει να υπάρχει ένα ενιαίο σημείο αναφοράς του καταναλωτή στην χώρα όπου υπάρχει το σύστημα αποζημίωσης. Το θέμα των συμψηφισμών επίσης είναι κάτι που πρέπει πολύ να κοιτάξουμε για να μην ε, γίνεται σε βάρος του καταθέτη. Εμεί πιστεύουμε ότι τέτοια μέτρα θα βοηθήσουν να υπάρχει αναγκαία εμπιστοσύνη του καταναλωτή στα συστήματα αυτά. Για το θέμα του συμψηφισμού στον Ηνωμένο Βασίλειο, πολλοί καταναλωτέ έχουν αποταμιεύσει και καταθέσει εκεί όπου έχουν και τι υποθήκε του. Κάτι το οποίο έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότεροι πάροχοι υποθηκών επιτρέπουν στου ε, ε, πελάτε του να έχουν και λογαριασμού ε, με καταθέσει. Η έρευνα έδειξε ότι η αρχή του ψηφισμού ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική για τους καταναλωτές και όσον αφορά τις υποθήκες ήταν κάτι που ξάφνιασε όλους όσους απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλουμε να, συ... να χρησιμοποιείται ο συμψηφισμό για τα συστήματα εγγύσεων καταθέσεων, για τη δημιουργία σύγχυση στους καταναλωτές, ε, χάνεται ρευστό καταθέσει των καταναλωτών και καθυστερούν και οι πληρωμές. Είχαμε πει για πέντε μέρες εργασίας, αλλά πέντε μέρες εργασίας είναι κάτι πολύ δύσκολο για τον καταναλωτή, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν ε, χαμηλά εισοδήματα και που χρησιμοποιούν τον προπολογισμό τους, ε, παίρνουν τα χρήματά τους δηλαδή κάθε εβδομάδα. Πληρώνονται κάθε εβδομάδα. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σύστημα στο οποίο έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές, που να είναι διάφανο, και βιώσιμο. Αν δεχτούμε ότι οι καταναλωτέ ε, λειτουργούν και αυτοί μέσα σε ένα πεδίο όλο και αυξανόμενων ε, ευθυνών προκειμένου να υπάρχει μια ασφάλεια στην αγορά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει προστασία για αυτούς. Και το σύστημα εγγύσεων καταθέσεων μπορεί να προσφέρει αυτή την προστασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα περνάμε στις Ιταλικές Συνεταιριστικές ε, Τράπεζες. Παρακαλώ. Κύριε κύριος σα σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε Βουλευτέ, θα ήθελα να σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας ε, παρουσιάσω το σύστημα εγγυήσεων των ε, αυστριακών συνεταιριστικών τραπεζών και τις επιπτώσεις της νέας ε, οδηγίας στο σύστημά μας. Εισαγωγικά ακούσατε ότι οι Ιταλικές συντριστικές τράπεζες δημιούργησε ένα νέο σύστημα για την εγγύηση των χρηματοπιστωτικών Ινστιτούτων και χαίρομαι που μπορούμε να σας βοηθήσουμε λιγάκι με τις εμπειρίες από την Αυστρία. Για τις αυστριακές συνεταιριστικές τράπεζες η μεταρρύθμιση της εγγύησης των αποταμιεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί το δικό μας συστήματα εγγύησης καλύπτει περισσότερο από την εγγύηση της αποταμίευσης. Η πελάτες μας καλύπτονται από ένα σύστημα πολλών επιπέδων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτή η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συστημάτων εγγύησης να μπορέσει να λειτουργήσει και στο μέλλον και να μην ε, περιοριστεί στο μέλλον μόνο για την εγγύηση των αποταμίευσεων. Αυτό ισχύει νομίζω για τις περισσότερες συνεταιριστικές ε, τράπεζες και τα ταμιευτήρια της Ευρώπης, γιατί όλα τα συστήματα εγγύησεως που προσφέρουν στον πελάτη μια ευρεία προστασία και δεν θα μπορεί με αυτή να αναποκριθεί ε, μια πρακτική ότι το ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους. Φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι στην Ιταλία και την Ισπανία επίση θα αναφερθούν στο σημείο αυτό. Επίση, είδαμε στο παρελθόν αυτό το σύστημα αποδείχτηκε πάρα πολύ θετικό στην πρόσφατη κρίση και γι' αυτό δεν θα πρέπει να θυσιαστεί στο βωμό μια οποιασδήποτε εναρμόνιση. Θεωρώ όμως ότι ακριβώς εδώ η πρόταση του εισηγητή κινείται οπωσδήποτε προς σωστή κατεύθυνση. Ορίζει ενιαίο επίπεδο προστασίας με κοινέ απαιτήσει με συγχωρείτε ε, το, ναι, το μικρόφωνο σας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η πρόταση του εισηγητή ορίζει ενιαίο επίπεδο προστασίας και κοινέ απαιτήσει επιτρέπει όμως διάφορες επιλογές για την επίτευξη του στόχου. Αυτή η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη την ποικιλομοφία στην ευρωπαϊκή αγορά τραπεζών πολύ καλύτερα από την πρόταση της Κομισιόν. Θα ήταν πραγματικά ε, πάρα πολύ άσχημο όλα τα συστήματα να περιοριστούν σε μια καθαρά λειτουργία paybox, αμυγούς εκμεταμίευσης, και έτσι θα μειώνεται το επίπεδο της προστασίας σε πολλά κράτη. Πώς ε, διαμορφώνεται το δικό μας σύστημα, το οποίο νηθήτησαν εν μέρη οι Ιταλοί οι συνάδελφοι, το κεντρικό σημείο είναι η συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης κινδύνου των ε, Ινστιτούτων του δικού μας τομέα. Μόνο έτσι μπορούν γλίγορα να ανοιχτευτούν καταστάσεις κρίσης και να υιοθετηθούν έγκαιρα αντίμετρα. Εάν χρειάζεται, οι άλλες ε, τράπεζες του τομέα διαθέτουν οικονομικούς πόρους για την εξυγίαση της κατάστασης αυτής της κρίσης. Μέχρι στιγμής αυτά τα μέτρα πρόληψης οδήγησαν πάντα στον στόχο τους και μπορούμε να πούμε πραγματικά ότι στα 120 χρόνια από τότε που ιδρυθήκαμε δεν υπήρξε ποτέ πτώχευση μιας ενδεστικής τράπεζας στην Αυστρία. Εάν παρόλα αυτά υπάρξει κάποια στιγμή μία πρόχευση, το, συστήματο, το σύστημά μας εγγυάται απόλυτα τις αποταμιεύσεις. Εκτός αυτού, οι τράπεζες μας υπόσχονται να προστατεύσουν και εκείνους τους ε, ε πελάτες που δεν καλύπτονται από τη νέα οδηγία της προστασίας των αποταμιεύσεων. Μπορεί λοιπόν ο πελάτη να βασιστεί απόλυτα στην προστασία μιας μεγάλης ομάδας, ενό μεγάλου ομίλου τραπεζών. Θα ήθελα όμω να τονίσω ότι αυτό μπορεί να το υποσχεθούμε μόνο εάν υπάρχει μια ολόκληρη ε, ομάδα διαφορετικών συστημάτων και ε, συστημάτων συγγνώμη, εγγύησης. Ε, είναι πολύ καλύτερο το δικό μας το σύστημα και αυτό που χρησιμοποιείται και στη Γερμανία της έγκαιρης παρακολούθησης και όχι της αντίδρασης στην περίπτωση πτώχευσης. Και επίσης ε, απαιτεί και λιγότερους πόρους. Η σταθερότητα, για τη σταθερότητα της ε, αγοράς τραπεζών είναι επίσης προτιμούμενη η εξυγένση γιατί παραμένει η εμπιστοσύνη των αποταμιευτών και δεν ανησυχούν οι καταναλωτές λόγω αντικών δημοσίευσεων στον τύπο. Ας μου επιτρέψετε να αναφερθώ στα κύρια σημεία της οδηγίας. Όσον αφορά την πρώτη διατύπωση της Κομισιόν, πραγματικά είχαμε σοκαριστεί. Γιατί όπως είπαμε αρνο, αγνοεί και αρνείται την πυκλομορφία των εθνικών αγορών τραπεζών. Όλα τα συστήματα περιορίζονται σε μια λειτουργία paybox Πραγματικά στην αρχή δεν κατάλαβα γιατί η Κομισιόν υπέβαλε αυτή την πρόταση. Μετά διάβασα όμως την αιτιολογική σκέψη 11, όπου η Κομισιόν λέει ότι σε περιπτώσεις, σε περιόδους κρίσης, οι ε, πελάτες προτιμούν τις ασφαλείς τράπεζες. Ε, γιατί όμως, τι είναι το κακό, είναι θέμα εμπιστοσύνης οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές γιατί στο παρελθόν απεδείχθησαν συχνά εκείνοι που προσπαθούσαν να, να ε, προσφέρουν κακώς εννοούμενα υψηλότερα επιτόκια, πράγμα που δεν ήταν προς του πελάτη, όπως το είδαμε και στις τράπεζες από την Ισλανδία και όχι μόνο εκεί. Όσον αφορά το ύψος του Ταμείου για την εγγύησει, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πολλές χώρες θα πρέπει να, προ... να δημιουργήσουν τώρα αυτά τα ταμεία εξάντε. Και είναι μεγάλη πρόκληση για εκείνους που μέχρι στιγμής είχαν ένα σύστημα εξπόστ. Επίσης ε, προβλέπεται να υπάρχει συμφωνία με το λεγόμενο Ταμείο Resolution Fund. Από δική μας ε, σκοπιάς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν μεγάλες μεταβατικές περιόδοι όπως το βλέπει και ο εισηγητής και μείωση του ύψους του ταμείου αυτού στο 1% ασφαλισμένων αποταμιεύσεων. Επίσης θα πρέπει να είναι δυνατόν ένα μεγάλο τμήμα του ταμείου να καλύπτεται με εγγύησεις για να μπορέσει ένα μεγάλο ποσοστό των ε, επενδύσεων να είναι διαθέσιμο. Και η ομάδα εργασία του Συμβουλίου υιοθέτησε ήδη μια σχετική πρόταση από την Πορτογαλία. Ένα κεντρικό θέμα είναι η χρήση των πόρων. Και εδώ προτείνει ρεαλιστικό και πραγματιστικό ε, τρόπο ο εισηγητής για να μπορέσει να προχωρήσει το σύστημα. Σύμφωνα με την τροπολογία του, ένα τρίτο του ταμείου θα πρέπει να χρησιμοποιείται για προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί δηλαδή η πτώχευση. Ορισμένοι λένε ότι μια τράπεζα θα προτιμήσει ο, ο ανταγωνιστής να πτωχεύσει παρά να τον βοηθήσει. Αλλά έχω να σας πω ότι στην πράξη στην Αυστρία βλέπουμε ότι μια τέτοια εξυγίανση είναι ληστική. και όχι μόνο σε ένα αποκεντρωμένο τομέα. Οι αυστριακές τράπεζες τα τελευταία χρόνια με την Bavac και την Κωνσταντσία Bank ε, έσωσαν δύο ανταγωνιστές εργαζόμενοι από κοινού γιατί ακριβώς αναγνώρισαν ότι το πλήγμα από μία πτώχευση θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Όσον αφορά τις προθεσμίες ε, αποζημίωσης, η Κομισιόν προτείνει 7 μέρες, μείωση σε 7 μέρες. Αυτό από σκοπιάς δικής μας δεν είναι ρεαλιστικό, γιατί είναι αδύνατον να μπορούν να εξεταστούν όλοι οι δικαιούχοι. Για σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολλοί ε, με δικαίωμα υπογραφή σε ένα ε, λογαριασμό. Αν το πληρωθούν τα χρήματα αυτά σε κάποιον που δεν τα δικαιούται, θα πρέπει μετά να τα ξαναζητάει πίσω το Ταμείο Εγγύησης. Και αυτό θα είναι ίσως εις βάρος των άλλων ε, ταμιευτών και επενδυτών. Επίσης, ο εισηγητής ε, προτείνει 5.000 ευρώ να καταβάλλονται σε 5 μέρες. Για λόγους ε, κοινωνικούς αυτό είναι κατανοητό. Το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να παραμένει ότι μπορεί η αποζημίωση αυτή να δοθεί σε έναν μη δικαιούχο. Θα ήθελα να μου τρεψετε στο τέλος να αφαιρθώ και σε μια πρόταση που, που εβάλαμε στις τελευταίες ε, συζητήσεις. Δηλαδή μια λεγόμενη co-insurance, ίδια συμβολή, ίδια συμμετοχή, που θα οδηγούσε στην ε, αναγνώριση του κινδύνου από τον ε, πελάτη. Γιατί αλλιώς ε, τα, οι πελάτες θα έδιναν τα χρήματά σου στην τράπεζα που προτείνει τα υψηλότερα επιτόχια, που καλό είναι εάν αυτό θα οδηγήσει στην επόμενη πτώχευση. Θα ήταν λοιπόν καλό να υπάρχει μια ίδια συμμετοχή και αυτό θα τέριαζε και στις προσπάθειες της Κομισιόν να αυξήσει την οικονομική παιδεία, όπως λέγεται, των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Αναγνωρίσαμε όμως ότι τις τελευταίες εβδομάδες ότι σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να επιτευχθεί πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ για προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή για οποιαδήποτε ερώτηση. Uh, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεντερίκο Κορνέλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εξ ονόματος ε, των, ε, <clears throat> της ε, συνεταιριστικής πίστης στην Ιταλία. Σας χαιρετώ. Έχουμε 420 περίπου μικρές και πολύ μικρές τράπεζες. Όλοι είναι στην τρίτη, η τρίτη εθνική ομάδα τραπεζών. Δεν είμαστε στο χρηματιστήριο. Πολύ μικρές τράπεζες. Το καταστατικό της ορίζει να βοηθήσουν την τοπική κοινότητα κάθε φορά και αν έχουν κέρδος δεν το διανέμουν διότι το 60% επανεπενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία και πάει για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας. Δεν είμαστε στο χρηματιστήριο παραπάνω. Ό,τι bonus ε, options στα ομόλογα και άλλα προβλήματα που δημιουργούνται με το χρηματιστήριο σε μας δεν υπάρχουν. Οι εταίροι μας είναι και οι καταναλωτές οι ίδιοι. Γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε ένα σύστημα προστασίας που να προσφέρει και στον καταναλωτή, δηλαδή στους εταίρους μας, ευρεία προστασία και αναλύσαμε τους λόγους της κρίσης που είναι κυρίως τρεις. Πρώτον δεν υπάρχει έλεγχος για τη ρευστότητα στα χρόνια πριν την κρίση. ένα πρόβλημα της διακυβέρνησης, governance, στο σύστημα των τραπεζών και κάνουμε ένα σχέδιο με την μεγάλη, πολύτιμη βοήθεια της ε, Κεντρικής Τράπεζας στην Ιταλία για ένα σύστημα IPS, σύστημα θεσμικής εγγύησης, IPS, με βάση το άρθρο 80. Για το, το IPS, το ταμείο αυτό, προσφέρει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα, χρηματοπιστωτική μάλλον σταθερότητα και πλήρη προστασία του καταναλωτή. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε η κυρία Κοτρέλα και παραξενεύτηκα πολύ γιατί εμείς κινηθήκαμε προς την κατεύθυνση της πλήρους προστασίας του καταναλωτή. Παράδειγμα, διότι αυτή η νομοθεσία, αυτός οι κανόνες ας πούμε, που θεωρούμε σωστοί αν και ο Αυστριακός συνάδελφος επισήμενο ορισμένα εκκρεμή σημεία, απαιτείται αυτή η νομοθεσία και ρύθμιση, υπάρχει όμω κίνδυνο αποφυγής. Και μιλάω ω τραπεζίτη αυτή τη στιγμή. Το έμεσο κόστος που συνδέεται με αυτό το 1% που πρέπει εκ των προτέρων να ε, καταβληθεί ω αφορά ε, καταθέσεις, μπορεί να υποχρεώσει τον τραπεζίτη να κινηθεί για αποφυγή. Δηλαδή, μπορεί να προσφέρει για ποσά ας πούμε 20, 30, 40 ευρώ μία αυτόματη μετατροπή σε άλλα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Εγώ είμαι απλός πελάτης μιας τράπεζας. Μέχρι τις 20-30 ευρώ μου φωνάζουν κοίταξε σου δίνω ένα ομόλογο, ένα άλλο εργαλείο μέσο χρηματοπιστωτικό με σεβασμό των MIFID, με σεβασμό της επιλογής μου αλλά τι κάνει ο τραπεζίτης. Μειώνει έτσι, συμπιέζει το έμεσο κόστος σχετικά με την εγγύηση και αποφεύγει, είναι εύκολο να το κάνει αυτό, αποφεύγει εντελώ το, το δικό σας σχέδιο. Αυτό είναι κίνδυνος, διότι de facto η φορολογητέα βάση εξαφανίζεται και λίγο το σύστημα αυτό δημιουργεί αυτό το μεγάλο κίνδυνο. Δεύτερος κίνδυνος, και μιλά πάλι ο τραπεζίτης, μείωση της ρευστότητα στην διατραπεζική αγορά. Διότι η ρευστότητα κατατίθεται στην ευρωαγορά. Και αυτή η ρευστότητα, αν μειωθεί, θα ανεβάσει το Euribor. Και η προστασία του καταναλωτή θα μεταφέρει αυτό το κόστος στα δάνεια, στο κόστος χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στον καταναλωτή. Πώς μπορεί να αποφευθεί η αποφυγή της εφαρμογής της τήρησης αυτής της νομοθεσίας. Εμείς έχουμε ένα δικό μας σύστημα εγγύσεων που προτείνουμε που εγγυράται όλα τα στοιχεία παθητικού, όχι μόνο τις καταθέσεις μέχρι 100.000. Εγγυάται όλα τα πάντα και το ποσό πάνω από τις 100.000 μέχρι 1 εκατομμύριο, ναι, μέχρι 2 εκατομμύρια, ναι. Και τα ομόλογα που βγάζει η τράπεζα και οποιοδήποτε άλλο εργαλείο χρησιμοποιεί. Βέβαια, για να έχουμε σταθερότητα απαιτούνται μέτρα για καλή διαχείριση της τράπεζας. Και το IPS, το δικό μας Ιταλικό Ταμείο, ασκεί ελέγχους με βάση τα νούμερα της τράπεζας, τη ρευστότητά της. Κάθε εβδομάδα ελέγχουμε τη ρευστότητα και ή δυνατόν κάθε μέρα. Και έλεγχο στα συστήματα διαχείρισης της τράπεζας, στο corporate governance της τράπεζας, διότι εκεί, από εκεί ξεκίνησε η κρίση ας πούμε, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κοιτάμε να δούμε, δουλεύει καλά. Κρύβει χαρτιά, τυχόν, το συνδικαλιστικό όργανο της τράπεζας δουλεύει σωστά, περιοδικά γίνεται αυτός ο έλεγχος. Τι πλεονεκτήματα μας δίνει αυτό το σύστημα. Ο καταναλωτής, αν εγγραφεί σε οποιαδήποτε προϊόν ή κατάθεση, να αφήσει ποσά πάνω από 100.000 ευρώ, ξέρει ότι η τράπεζα, η συνεταιριστική τράπεζα στην περίπτωση αυτή, είναι υπό την επαγρύπνηση και της Κεντρικής Τράπεζας στην Ιταλία και από το δικό μας Ταμείο Εγγύησης, όπου όλες οι τράπεζες έχουν δώσει ένα τμήμα εξουσιών ως ένα τρίτο πρόσωπο και έρχεται και κάνει έλεγχο. Αυτό είναι σημαντικό διότι δημιουργείται στον καταναλωτή μία εκ των προτέρων προστασία. Σταθεροποιείται η τράπεζα, αποφεύγεται η χρεοκοπία. Ενισχύεται η εμπιστοσύνη. Γιατί ακόμα κι αν ο τραπεζίτης μετατρέψει το ενεργητικό παθητικό με τρόπο που να αποφύγει την νομοθεσία και σε βάζει να πάρεις ομόλογα ή άλλου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία αντί για καταθέσεις, εμείς έτσι κι αλλιώς όλα τα προστατεύουμε. Ενώ με το DGS είναι εκτός προστασίας. Με βάση όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σταθερή εποπτεία, μόνιμη εποπτεία. Η πρότασή μας είναι να ευνοηθούν αυτά τα εργαλεία που θα αυξήσουν την προστασία του καταναλωτού και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και για το άρθρο 11 της πρότασης, το IPS θα έχει μεγαλύτερη κάλυψη από το 65% περίπου που προβλέπει η πρόταση. Ανώτερο γιατί? Διότι έχουμε έλεγχο μόνο για το IPS έλεγχο ρευστότητας και του corporate governance με μεγαλύτερη προστασία για τον καταναλωτή. Αυτό είναι το αίτημά μας. Να έχουμε μία κάλυψη 100%. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, συμφωνούμε με αυτά που είπε ο Αυστριακός συνάδελφος και συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω ένα σημαντικό. Η εποπτεία, η πρόληψη και η δυνατότητα παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μικρών τραπεζών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από τις Βρυξέλλες ή από το Λονδίνο για μια μικρή τράπεζα στην Καλαβρία ή σε μια μικρή περιφέρεια της Βόρειας Ιταλίας. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε προληπτική δράση εξάντε εκ των προτέρων. Γιατί σε κάθε κρίση το συνεδριστικό κίνημα των τραπεζών στην Ιταλία δεν ζήτησε ούτε ένα ευρώ, ούτε μία λιρέτα από την κυβέρνηση. Λύσαμε, επιλύσαμε όλες τις κρίσεις μόνοι μας με το δικό μας σύστημα εγγύσεων, κάπως με αυτό, παρόμοιο με αυτό που κάνουν οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί συνάδελφοι, να προστατεύσουμε την αυτονομία μας και το θεωρούμε σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you um, Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα περνάμε στον ε, Λουίς Τεχέρο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Λουίς Τεχέρο και είμαι επικεφαλής ε, των πολιτικών για την ρύθμιση της, ε, του Ισπανικού, της Ισπανικής Αποταμιατικής Τράπεζας. Θα σας πω πώς έχει κατάσταση στην ισπανική αγορά. Εμείς πιστεύουμε ότι κάνουμε πολλά από αυτά που περιλαμβάνονται στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως για παράδειγμα και στην πρόταση του συγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης χρησιμοποιούμε και μηχανισμούς που δεν είναι υποχρεωτικοί προς το παρόν, αλλά οι οποίοι αποτελούν ένα πλαίσιο υπέρ της οικονομικής σταθερότητας, αλλά περιλαμβάνουν και την ελαστικότητα, την ευελιξία, για να μπορούμε και προληπτικά, αλλά και διορθωτικά μετά, να μας ε, βοηθήσουν σε περίπτωση οικονομικών κρίσεων. Θα σας πω ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ισπανικού συστήματος ταμιευτηρίων. Καταρχήν, όλα τα πιστοτικά ιδρύματα, όλα τα δαμευτήρια πρέπει να συμμετέχουν σε ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Και γι' αυτό και δημιουργήθηκαν τρία διαφορετικά ταμεία, ένα για τις τράπεζες, ένα άλλο για τα ταμιευτήρια και ένα τρίτο για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν καλύπτονται μόνο οι καταθέσεις αλλά και οι τίτλοι που έχουν κατατεθεί στην ε, τράπεζα. Αλλά δεν ε, έχουν εκδοθεί από την ίδια. Δεν καλύπτονται καταθέσεις ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του δημόσιου τομέα ή εταιριών. Ούτε καλύπτονται και ορισμένα ειδικά πράγματα όπως είναι τα πιστοποιητικά καταθέσεων ή τα δευτερεύοντα χρέη ρέπος κλπ. Αυτά δεν καλύπτονται. Έρχομαι τώρα στα χαρακτηριστικά. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε είναι ότι τα τρία συστήματα αφορούν ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, είναι εντελώ χωριστά τα συστήματα αυτά από αυτούς που δίνουν τα χρήματα, είτε πρόκειται για το κράτος, είτε πρόκειται για κάτι άλλο. Είναι δηλαδή ένα σύστημα εντελώς διακριτό, χωριστό, που χρησιμοποιεί ενεργητικό υψηλής ποιότητας και πρόκειται για συστήματα που χρηματοδοτούν 100% εξάντε και που καλύπτουν έναν στόχο 1% για τα, τις καταθέσεις που καλύπτονται. Εδώ είναι η πρόταση και της οδηγίας, έτσι, που λέει να είναι 1,5%. Εδώ ίσως δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι το 1% φτάνει και όσον αφορά τώρα τους τίτλους, υπάρχει μια κάλυψη 5% για τους τίτλους οι οποίοι βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση για την εισαγωγή και 5% για τους άλλους τίτλους. Αν καλύπτεται ο στόχος, μπορούν να δοθούν, να ζητηθούν μάλλον και χαμηλότερα επίπεδα αλλά περισσότερα εφόσον το σύστημα, επειδή προέκυψε κάποιο έκτακτο γεγονός, δεν έχει απόθεμα. Τέλος, προβλέπεται και δυνατότητα η ίδια η Τράπεζα της Ισπανίας να μπορεί να παρέμβει, εφόσον χρειαστεί σε έκτακτες περιπτώσεις. Και έρχομαι τώρα στο πιο ενδιαφέρον, πιστεύω, που είναι πόσο χρησιμοποιείται το σύστημα εγγύσεων καταθέσεων στην ισπανική αγορά. Με δύο τρόπους. Πρώτον, στόχος είναι, ο συνήθις στόχος, να καλυφθούν οι καταθέτες. Με στόχους που ορίζουμε και εφόσον πραγματοποιηθούν ξεκινάει η πληρωμή των καταθετών και οι πληρωμές εφόσον αποφασιστεί η πληρωμή, γίνεται το πολύ σε 20 εργάσιμες ημέρες. Από τη στιγμή δηλαδή που είτε η Τράπεζα της Ισπανίας ή κάποιο δικαστήριο πάρει την απόφαση για αποζημίωση των καταθετών. Κάτι άλλο ενδιαφέρον πιστεύω εδώ, όπου διαφοροποιούμαστε κάπως από τόσα λέει η οδηγία, είναι το εξής. 20 εργάσιμες μέρες για μας είναι μια λογική προθεσμία. Το να μιλάμε για πέντε μέρες, αυτό σημαίνει σε πολλές περιπτώσεις μεγάλες ε, δυσκολίες για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου στόχου, λειτουργικής φύσεως. Αυτά όσον αφορά τη συνηθισμένη χρήση του συστήματος εγγύσεων καταθέσεων. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη πτυχή εδώ, ένα δεύτερο είδος χρήσης του συστήματος αυτού και είναι η επίλυση τραπεζικών ε, κρίσεων. Το σύστημα προβλέπει στην Ισπανία, προβλέπει να διοθετούνται μέτρα ώστε προληπτικά να μπορούμε να αποφύγουμε αποζημιώσεις στους καταθέτες. Και έτσι προστατεύουμε και τα 100.000 των ε, καταθετών, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, όπως καταλαβαίνετε εφόσον προλαμβάνουμε τη ζημιά. Πρόκειται λοιπόν για μέτρα είτε καθαρά προληπτικά, όπου το σύστημα εγγύσεων καταθέσεων πληρώνει το κεφάλαιο αυτού που ζητάει τη βοήθεια, είτε για ζημίες, είτε για δάνεια, είτε για εγγύησεις, είτε για άλλου είδους πρωτοβουλίες, όπου προληπτικά αποφεύγεται να μπει το Ίδρυμα σε δυσκολίες. Στη συνέχεια έχουμε μέτρα αναδιάρθρωσης, μέτρα εξυγίανσης του οργανισμού. Πολλές φορές διευκολύνεται η αγορά από κάποιον ανταγωνιστή ή μιλάμε για συγχώνευση. Έτσι υπάρχει εγγύηση μέρους των καταθέσεων και μεταφέρεται το ενεργητικό αλλού κλπ. Τέλος υπάρχει και δυνατότητα να ζητήσει η Τράπεζα της Ισπανίας μέτρα σχετικά με την διαχείριση των χρηματοπιστωτικών ιδρωμάτων και μπορεί να υπάρχει θέμα βελτίωσης των εσωτερικών ελέγχων ή να υπάρχει βελτίωσης της διαχείρισης του κινδύνου. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο διπλός στόχος καλύπτει τα όσα ζητάει η οδηγία. Είναι δηλαδή η δυνατότητα το Ταμείο Εξυγίανσης το οποίο δημιουργείται χρησιμοποιείται για να προστατεύσει τις καταθέσεις. Τέτοιου είδους μέτρα για μας είναι πολύ σημαντικά διότι σαν κύριο πλεονέκτημα έχουν την ελαστικότητα. Ελαστικότητα στην διαχείριση σε περίπτωση τραπεζικής κρίσης. Η ελαστικότητα αυτή, η ευελιξία αυτή που προσφέρεται στον επιθεωρητή να επιλέξει το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να προστατεύει καλύτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο καλύτερος τρόπος για την προστασία των πόρων και τελικά καταλήγουμε σε καλύτερη χρήση των πόρων αυτών. Τέλος, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην τρέχουσα κρίση, το σύστημα εγγύσεων καταθέσεων του Ισπανικού Ταμιευτηρίου βοήθησε να προστατεύσουμε έτσι το ταμιευτήριο της Καστίγια Λαμάντσα. Με την ε, απόκτηση προτιμησιακών συμμετοχών για ένα δις 300 εκατομμύρια ευρώ. Είναι προφανές ότι οποιοδήποτε σύστημα εγγύσεων καταθέσεων ταμιευτηρίων και αν έχουμε, δύσκολα θα φτάνει σε περίπτωση συστημικής κρίσης, αν και αυτήν που έχουμε. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι πέρα από το καθορισμό των γενικών χαρακτηριστικών των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων πρέπει να δούμε λίγο και τα προληπτικά μέτρα τα οποία θα προλάβουν μια παρόμοια κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much and many Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που τήρησαν και χρόνο τους μπορούμε να περάσουμε στις των βουλευτών και θα ήθελα καταρχήν να στραφώ στον τον Πίτερ Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλήσαντες όχι μόνο επειδή δέχονται θετικά ορισμένε πτυχές της εκθέσή μου αλλά και γιατί μας έδωσαν μια πολύ ωραία εικόνα της κατάστασης στις χώρες αυτές. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα αναφερθώ στα σημεία που ε, συμφωνείτε, στα οποία συμφωνείτε μαζί μου, αλλά εκεί που υπήρχαν επικρίσεις να σας πω γιατί υποβάλλω την πρόταση συγκεκριμένα που μου φαίνεται σωστή. Καταρχήν, εξετάσει κατά πόσο εγγυήσεις θα πρέπει να θεωρηθούν ταμιεύσεις ε, ή μάλλον εισφορές ε, στο Ταμείο εγγύησης; Εγώ δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο γιατί νομίζω ότι μόνο μια πραγματική πληρωμή καταβολή εξάντε μπορεί να βοηθήσει γιατί αυτή λειτουργεί αντικυκλικά. Η ενώ μια εγγύηση κατά τη γνώμη μου είναι μια και καλυμμένη εξ χρηματοδότηση. Το 1,5% σαν στόχο μου φαίνεται ότι η λύση που προτείνεται ε, λαμβάνει υπόψη αυτά που θέλετε. Προβλέπετε μια ε, σωστή ετήσια επιβάρηση των επιχειρήσεων με αυτό που προτείνουμε εμείς είναι το ίδιο όπως αν έχουμε 1% στα 10 χρόνια, αλλά ε, εμείς προτείνουμε 15 χρόνια, μακρύτερο χρονικό διάστημα, την ίδια επιβάρυνση όμως. Όσον αφορά τις ε, προθεσμίες αποζημίωσης και το ότι μπορεί να καταβληθούν τα χρήματα αυτά χρεωσίτως σε κάποιον που δεν τα δικαιούται. Εγώ ομολογώ ότι δεν κατανοώ το πρόβλημα. Εάν έχουμε μια λειτουργούσα τράπεζα και υπάρχουν πολλοί δικαιούχοι που μπορούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον να αδειάσουν, το, ε, αδειάσουν αυτό το λογαριασμό, πού είναι η διαφορά αν πτωχεύσει μια τράπεζα και συμβεί ακριβώς το ίδιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι προβληματικό. Όσον αφορά την ίδια συμμετοχή των πολιτών, αυτή η σκέψη της υπεύθυνη επένδυσης μπορώ να τη συμπεριστώ. Από την άλλη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλοί πολίτες ε, δεν μπορούν να κατανοήσουν πραγματικά ποια είναι η συμπεριφορά της τράπεζάς τους κατά πόσον αυτή η τράπεζα στην οποία πηγαίνουν τα χρήματά τους ε, είναι μία που έχει ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο. Ξεπερνάμε νομίζω εδώ τις δυνατότητες του πολίτη και δημιουργούμε χαμηλότερη προστασία του καταναλωτή. Το θέμα των 20 ημερών, κατά πώς θα το διατηρήσουμε ή όχι. Εγώ προτείνω ή 20 μέρες, αλλά στις πρώτες 5 μέρες να πληρωθούν γρήγορα 5.000 ε, ευρώ στον πολίτη. Αυτό λαμβάνει υπόψη και τις δύο πτυχές. Και τη σκέψη που έχετε εσείς ότι δεν επιτρέπεται να υποσχεθώ οτιδήποτε όσον αφορά τις προθεσμίες αυτές τις αποζημίωσεις που δεν μπορώ να τηρήσω και με το να μην τηρηθούν οι προθεσμίες αυτές να καταστρέψουμε την εμπιστοσύνη των ε, πολιτών. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ στην ε, ε, Ήπειρό μας ε, δεν μπορούν να επιζήσουν 20 μέρες χωρίς καθόλου χρήματα και χωρίς δυνατότητα να αποσύρουν χρήματα. Και γι' αυτό νομίζουμε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη μας και να φροντίσουμε πιο εύκολα και πιο γλίγορα να επανέλθουν σε μια κατάσταση ρευστότητας οι ε, καταναλωτές. Μετά, το θέμα της επιβάρυνσης των ε, χρηματοπιστωτικών ε, Ινστιτούτων με την ε, υποχρέωση καταβολής στα συστήματα εγγύησης. Και αν γι' αυτό οι, οι τράπεζες περνάνε σε άλλα προϊόντα που δεν καλύπτονται, όπως είπε ο Σκονέλη. Τρία πράγματα. Είναι θέμα από απόφαση του καταναλωτή κατά πόσον ε, παιδί τα χρήματά του στο ταμιευτήριο που λέει ότι εντάξει δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο και χαμηλή, ε, ε χαμηλή τόκηση και από την άλλη μεριά το δίνει κάπου αλλού που έχει περισσότερες ε, δυνατότητες ε, κέρδους. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε βάσει της ε, Βασιλείας 3 ότι μια τράπεζα δεν θα πέναγε γι' αυτό σε έναν τομέα που είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Επίσης θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η συμβολή της τράπεζας όσον αφορά τα συστήματα εγγύησης των αποταμιεύσεων εξαρτάται από πόσο ε, επικίνδυνη είναι η συμπεριφορά επένδυσης μιας τράπεζας. Αν δηλαδή μία τράπεζα θέλει να περάσει από μία ασφαλή συμπεριφορά σε μία πιο επικίνδυνη, αυτό έχει και επιπτώσεις στην ε, συμβολή της τράπεζας αυτάς. Γι' αυτό θα ήθελα να βάλω ένα ερωτηματικό κατά πόσο ε, μπορεί να υπήρχε εδώ ε, ο κίνδυνος να περάσουν οι τράπεζες σε πιο επικίνδυνα προϊόντα. Γι' αυτό το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτό μάλλον συζήτησα δεν ήταν ερώτηση. Και θα περάσω στους άλλους βουλευτές νομίζω πριν επανέλθω στο πάνελ των ομιλητών. Η Βίκη. Um, Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε για τα διάφορα αυτά συστήματα στις διάφορες χώρες, πώς λειτουργούν, την εμπειρία σας πριν και μετά την κρίση και να μην ξεχνάμε τα πάρα πολλά μικρά ιδρύματα που διαχειρίζονται καταθέσεις και δάνεια. Για να καταλάβω κάτι, πώς δουλεύει το σύστημα αμοιβαίας εγγύησης. Η Γερμανία και η Αυστρία το ανάφερε. γιατί μπορεί να έχουμε ε, ένα είδος ε, αποτέλεσμα ντόμινο. Αν το σύστημα αμοιβαίας εγγύησης σημαίνει ότι κάθε πιστοτικό ίδρυμα είναι υπόλογο και για τις καταθέσεις μέχρι ένα ορισμένο ποσό αλλά και για επιπλέον κεφάλαιο και ρευστότητα αν κάπου το σύστημα καταρρεύσει. Ή μιλάμε για διαφορετικό κίνδυνο από ό,τι μιλάμε όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή. Γιατί αν δούμε το, από τη, σκοπιά του CRD, αυτές οι αμοιβέ εγγύησει δεν ε, ε, βάζουν κεφάλαιο παράλληλα για κάλυψη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι κάνετε εσείς ως επιμέρους ιδρύματα έτσι ώστε να υπάρχει επαρκές κεφάλαιο για το ενδεχόμενο αυτό χρέος και κίνδυνο προκειμένου να σταματήσει αυτό το η δράση ντόμινο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Θέλω μια πληροφορία για την πρόταση του Πίτερ Ζήμον σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν στα προγράμματα εγγύησεων που έχετε Ποιος είναι ο δείκτης προστασίας σε σχέση με τις διάφορες προτάσεις. Πόσο κεφάλαιο πρέπει να βάλετε στην άκρη, ανάλογα με την κάθε πρόταση. Και τι διαφορά υπάρχει από χώρα σε χώρα. Γιατί μπορεί να έχει μια χώρα που να έχουν πιο ψηλό προφίλ κινδύνου, άλλου πιο χαμηλό. Οπότε η πρόταση είναι και αυτή διαφορετική. Το συνολικό ποσό που θα βάλετε στην πάντα θα αυξηθεί ή θα μειωθεί και πόσο μεγάλη είναι η διαφορά αυτή. Μια ερώτηση για τον κύριο Κουπάη. Συναντηθήκαμε και συζητήσαμε και στο παρελθόν και ξέρω ότι είσαι άνθρωπος με πολλές ικανότητες. Θέλω λοιπόν να καταλάβω, εσείς τι ρόλο παίζετε. Από τη μια μεριά έχετε, είστε, είστε αυτός ο οποίος ε, εισήγαγε το έφτη και ταυτόχρονα δουλεύετε για τη γερμανική κυβέρνηση. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων εδώ ή όχι. Γιατί εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ σε μεγάλο ποσοστό να συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις του συναδέλφου Σίμων. Θα υποστηρίζω μάλιστα. Ίδιος το θέμα τη ανοιχτή της ανοιχτής, ε, των τραπεζών που μας ενδιαφέρει και εμάς. Έχω μια ερώτηση προς τους υπερογνώμονες. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ορισμένε χώρες που συνεργάζονται μαζί μας σε ένα νομικό πλαίσιο, όπως παραδείγματος χάρη Νορβηγία, χώρες δηλαδή που έχουν υψηλότερα εγγυημένα ποσά. Ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές ε, σκεφτήκαν πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση γι' αυτό. Γιατί τα χρήματα αυτά στην Ευρώπη βέβαια ε, μπορούν πολύ γλίγορα να κυκλοφορήσουν και να αποσταλούν από εδώ και εκεί. Υπάρχουν συγκεκριμένε παρατηρήσει ή συστάσει που θα μπορούσατε να μα κάνετε εσεί ω συζητητέ. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Θα έλεγα να επανέλθουμε στο πάνελ με τη σειρά με την οποία μίλησαν. Δύο λεπτά ο καθένα σύμφωνα με το χρόνο που έχουμε. Να παρεστείτε λοιπόν στι. Ε, Παρατηρήσει που σα ενέφερα περισσότερο και να απαντήσετε ίσω και σε κάποιες από τι ερωτήσει. Ίσως ε, ένα σχόλιο για την διπλή χρήση των ε, ποσών των ταμείων. Δηλαδή για τη διαχείριση χρήσης και για την εγγύηση της, ε, της κατάθεσης. Ο Τέικ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Κίπαρ, το οποίο ε, είπε ότι είμαι ιδρυτής ε, και αντιπρόεδρος του ΕΦΤΗ και αυτό είναι ο ρόλο μου εδώ. Οι θέσεις που παρουσίασα εδώ σήμερα είναι γραπτέ θέσει του Ευρωπαϊκού ε, Ταμείου αποταμίευσεων. Είπε ταυτόχρονα ότι είμαι και επίσημος συμπεριλαμβανόμενος για την γερμανική κυβέρνηση. Ε, αυτό δεν βλέπω να υπάρχει μια σύγκρουση. Γιατί εγώ εργάζομαι για τα συστήματα αυτά εγγυήσεων, από τα οποία αποκομίζω εμπειρογνωμοσύνη, τις εργασίες μου στις Επιτροπές για την Βασιλεία Επίσης αποκομίζω κάποια ε, στοιχεία εμπειρογνωμοσύνης τα οποία ε, ε, θεωρεί πάρα πολύ θετικά η γερμανική κυβέρνηση. Και υπάρχουν στην ομάδα αυτή, στην οποία συνεργάζομαι στην γερμανική κυβέρνηση και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις όταν έρχομαι κάπου να μιλήσω μιλάω εξονοπτός κάποιας από αυτές τις ε, οργανώσεις που εκπροσωπώ και εδώ σας είπα ξεκάθαρα ότι αυτά που σας είπα είναι θέσεις εύτη δεν είναι προσωπικές μου απόψεις, απόψεις της εύτη δεν υπάρχει καμία σύγκρουση και ό,τι και να κάνω οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ διαφανές. Δεν απέκρυψα τίποτα. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτός και σας λέω ακριβώς περί την σας πρόκειται. Επί τώρα. Ο κ. Σπάς αναφέρθηκε κατά πόσον η ψηλότερη προστασία σε ορισμένους χώρους μπορεί να είναι προβληματική. Στην έρευνα που έκανε η Κομισιόν το 2000 και το 2000 το σκεφτό υπήρχαν οι σκέψεις για την αρχή του λεγόμενου topping up και υπήρχε και απαγόρευση εξαγωγής, δηλαδή ήταν ε, ε, πολλές φορές υψηλότερο το επίπεδο προστασίας από την ε, χώρα που την προέρχονται παρά στην χώρα υποδοχής. Τώρα μας είπαμε ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει τέτοια στρέβλωση του ανταγωνισμού και γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η απογόρευση της εξαγωγής της προστασίας. Ξέρουμε περιπτώσεις στις οποίες θεωρητικά αυτή η διαφορά της εγγύησης οδήγησε σε μια απορρόφηση κεφαλαίων σε περιπτώσεις και εποχές κρίσης δηλαδή. Αλλά για δημοσιονομικέ κρίσει, βέβαια, δεν είναι το σωστό πλαίσιο αυτό. Χρειαζόμαστε διαφορετικό πλαίσιο για την προστασία αυτή. Εγώ προσωπικά ω εμπειρογνώμονα δεν βλέπω να υπάρχουν προβλήματα. Και μέσα στα πλαίσια της πρότασης της ε, Κομισιόν είναι όμω αντίθετο με την βασική ιδέα της αναρμόνισης για τις 100.000 ευρώ. όσον αφορά τα θέματα της ε, εγγύησης των Ινστιτούτων, των συστημάτων εγγύησης των Ινστιτούτων μάλλον, των χρηματοπιστικών Ινστιτούτων. Δεν θέλω να πω τίποτα γιατί εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονα σε αυτά. Και όσον αφορά μια παρατήρηση του κυρίου Σίμων, 1% σε 10 χρόνια ή 1,5% σε 15 χρόνια δεν τίθεται μόνο το θέμα της αιτήσιας χρηματοδότησης αλλά και της σχετικότητας. Και εξετάζουμε κατά πόσο αυτό χρειάζεται, γιατί η σχετικότητα σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης. Για το 1,5% έχουμε αμφιβολίες, γιατί με δύο εξαιρέσεις στην ε, ε, χρηματοπιστωτική κρίση στην Ισλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή μέσω των Ισλανδικών τραπεζών, δεν υπήρχε ανάγκη ποτέ για κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, και το πόσο πολύπλοκο είναι. ας πούμε να αναφερθούμε σε κοινές, κοινούς λογαριασμούς ε, από συνειδιοκτήτες. Ε, καμιά φορά δεν υπάρχει δυνατότητα κατανόηση. Ευχαριστώ. Υπάρχουν και άλλοι ομιλητές μετά από εσά. Με συγχωρείτε θα σας διακόψω. Ωραία. Ωραία. Τελευταία παρατήρηση για την ίδια συμμετοχή, συμβολή, συμμετοχή. Το καταργεί η Κομισιόν, δεν το εισαγάγει στην έκθεσή τη και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό είναι και τμήμα τη Επιτροπή Βασιλεία ότι δεν θα πρέπει να ισχύει αυτή η ίδια συμμετοχή για συστήματα αποταμίευση. Γιατί κάποιο που μπορεί να πάρει 100% ε, θα όπως είπε ο κύριος Σίμαν, δεν μπορεί ο καταναλωτής να κρίνει το πόσο επικίνδυνη είναι η μετάβαση στην οποία καθέτει τα χρήματά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσετε σε όλα και ότι πολύ θα θέλατε. Η ε, κυρία Κοτρέλα. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη για την χρηματοδότηση των αμοιβαίων εγγύσεων καταθέσεων δεν έχουμε κάτι τέτοιο, οπότε δεν θα μπορούσα να το σχολιάσω. Αλλά θα αναφερθώ σε άλλες χώρες, χρήματα τα οποία για παράδειγμα πήγαν στην ε, Ιρλανδία όταν έβαλε χωρίς οροφή όριο. Και Μιλήσαμε τότε για τον κίνδυνο, γιατί δεν υπήρχε προχρηματοδότηση του συστήματος, άρα δυνητικά υπήρχε κίνδυνος. Τα χρήματα δεν προστατεύονταν και εμείς λέμε στους καταναλωτές να το λαμβάνετε υπόψη σας, άμα θέλετε να βάλετε τα χρήματά σας σε έναν Ιρλανδικό λογαριασμό. Τι μπορεί να σημαίνει για σας αν υπάρξουν δυσκολίες στο συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αυτό ήταν το μόνο που είχα να πω. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ο επόμενο. Μα ε, ρωτήστε το, το τι εμπειρίε έχουμε από την κρίση. Εγώ δεν μπορώ να σα πω παρά τι έγινε στην Αυστρία και αναφέρθηκα σύντομα στην έκθεσή μου. Στην κρίση είχαμε δύο εκτόσει, η Μπάβακ και η Κωνσταντσια, αυτές οι δύο τράπεζε, όπου πραγματικά αντιμετωπίσαμε το θέμα ρεαλιστικά, υπολογίσαμε τι θα κόστιζε να αφήσουμε τι τράπεζε αυτέ να πτωχεύσουν και τι θα κόστιζε να τις εξηγιάνουμε. Και όλες οι αυστριακές τράπεζες από κοινού αποφάσισαν ότι τα μέτρα εξυγίανσης όχι μόνο θα ήταν οικονομικότερα και, αλλά και όσον αφορά την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα ήταν η καλύτερη λύση. Όσον αφορά την ε, ε, το φαινόμενο μπούμεραν. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν όρια μάλλον επιβάλληση των τραπεζών για τα οποία θα μπορέσουν να ε, επιβαρυνθούν. Κατόπιν αυτών υπάρχει ε, αυτό το φαινόμενο του ντόμινο. Βέβαια κάθε μέτρο δεν μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία. Ο εισηγητής ε, προβλέπει ένα όριο, δηλαδή ένα τρίτο του ταμείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξυγίανση. Εάν ξεπερνάμε το ποσοστό αυτό, είναι δυνατόν να γίνει μόνο με συνεργασία της ε, εποπτικής αρχής. Υπάρχει εδώ δηλαδή ένα όριο που μου φαίνεται ότι είναι μια λογική λύση. Και επαναλαμβάνω θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλο το θέμα της χρήσης των πόρων σε σχέση με το ταμείο αυτό σε αυτό το λεγόμενο Resolution Fund, θα πρέπει να εξασθούν από κοινού. Ξέρω ότι η Κομισιόν δεν έχει προχωρήσει σε αυτό όσο έχει προχωρήσει για την εγγύηση των καταθέσεων, αλλά έχω κάποια στοιχεία ότι θα μπορεί να εξασθεί αυτό από κοινού, ε, από την Κομισιόν, με τα δύο αυτά μάλλον από κοινού. Τελευταίο, ε, το θέμα της, ε, του κινδύνου ε, μπορούμε να αναφερθούμε σε πάρα πολλές ε, τράπεζες. Έχουμε 520 ε, τράπεζες και γι' αυτό ο κίνδυνος δεν είναι καθόλου περιορισμένος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, κύριος Κορνέλη. Ευχαριστώ. Θα προσθέσω να δώσω τρεις απαντήσεις στον κύριο Σίμων στην Βρετανή συνάδελφο και στο, στον Γκίκολτ, στον κύριο Σίμωνα. Η αποφυγή δεν καλύπτεται από την Βασιλεία, Ερώτηση. Ίσως δεν εκφράστηκα σωστά. Κάντε λάθος αν θεωρείτε ότι η Βασιλεία ζητάει σε περίπτωση αποφυγής μια στάθμιση μεγαλύτερη του κεφαλαίου. Διότι να περάσουμε από μια κατάθεση σε ομόλογο ή άλλο εργαλείο, είμαστε παραμένουμε στο παθητικό της ε, επιχείρησης, ενώ η Βασιλεία 2 ουσιαστικά προσπαθεί να στραφεί στα δάνεια που δίνει η τράπεζα, στα ενεργητικά στοιχεία της τράπεζας. Ένας λοιπόν τραπεζίτης που μεταθέτει από τις καταθέσεις προς άλλα εργαλεία δεν έχει αύξηση του κεφαλαίου του τυρ 1. Αποφεύγει όμως, αποφεύγει, ασκεί αποφυγή. Και έτσι ενθαρρύνεται αυτή η τάση. Τώρα απαντώ στην ε, ε, Βρετανίδα Ευρωβουλευτή. Πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα εγγύησης που ρωτήσατε. Οι τράπεζες συνήθω πτωχεύουν ε, λόγω, λόγω ρευστότητας. Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να σώσει το σύστημα. Ο πυλώνας λοιπόν ρευστότητα είναι πολύ σημαντικό και στην περίπτωσή μας εμείς ένα νούμερο θα σας δώσω. Ε, για μπορεί να μας ζητήσουν 5 εκατομμύρια με στατιστικές μεθόδους θα δώσουμε, ε, αν μας ζητήσει 500 εκατομμύρια θα δώσουμε πάνω από ένα δις. Πολύ μεγαλύτερη προστασία δηλαδή. Προληπτικά δρούμε, προληπτικά. Διότι αν δεν δράσουμε προληπτικά και αν δεν παρέμβουμε, όπως είπε και ο αυστριακός συνάδελφος, τα συστήματα αντιδρούν απλώς δεν υπάρχει μια πραγματική δυνατότητα υποστήριξη ακόμα και με τρίου μεγέθους σοκ, ενώ η προστασία που δίνει το σύστημα EPS, η Ιταλική εμπειρία, Γερμανική εμπειρία, η Αυστριακή εμπειρία το αποδεικνύει, προβλέπουμε μεσαίου μεγέθους σοκ. Και για τον κύριο Γκίγκολτ. Ποιο είναι το βάρος της εισαγωγής αυτής της νέας ρύθμισης νομοθεσίας. Το βάρος για μας που είμαστε μια κλασική τράπεζα είναι περίπου 400.000 ευρώ επιπλέον. Αυτή λοιπόν η νομοθεσία βαρύνει τις κλασικές τράπεζες βιοτεχνικού τύπου, ας πούμε, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, που θα χρηματοδοτήσουν, που χρηματοδοτούν μάλλον μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ λιγότερο επηρεάζει τις τράπεζες επενδύσεων που δεν το κάνουν αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Λουίτζι Φέρο. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάω από αυτό το τελευταίο σημείο. Εμείς δεν έχουμε εκτιμήσεις για το κεφάλαιο στον τραπεζικό τομέα πάντως της Ισπανίας και δεδομένου ότι ξεκινάμε από ένα εξάντε σύστημα εγγύσεων καταθάσεων, οι επιπτώσεις θα είναι εφόσον αυξηθεί κατά μισό της εκατό το ποσοστό και θα είναι παραπάνω εάν βασιζόμαστε σε eligible deposits αντί για covered deposits. Η επίπτωση θα είναι μικρότερη σε εμά από τις άλλες χώρες όπου δεν υπάρχει τέτοια εξάντα κεφαλοποίηση. Όσον αφορά τώρα την ε, δυνατότητα διαφυγής κεφαλαίου σε άλλες χώρες, εμείς πιστεύουμε ότι με το σημερινό επίπεδο κάλυψης 100.000 ευρώ και πάντα μιλώντας για τα ταμιευτήρια, το επίπεδο αυτό καλύπτει ένα πολύ ψηλό ποσοστό των καταθετών. Άρα η δυνατότητα να υπάρξει αυτή η διαφυγή κεφαλαίου θα είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας για τη συμμετοχή σας εδώ. Έτσι ολοκληρώνεται η ακρόασή μας. Ευχαριστώ όλους σας. Στα μέλη της Επιτροπής μας λέω ραντεβού όχι στις 3, στις 2, γιατί έχουμε τον Κάρι Γκένσλερ, ε? μην το ξεχνάτε. 2 η ώρα, όχι στις 3, 2 η ώρα εδώ. Είναι ανοιχτή συνεδρίαση και για άλλους όποιος θέλει μπορεί να έρθει.